για... Καλησπέρα σας. Θα συνεχίσουμε με την ημερήσια μας διάταξη. Έχουμε να συζητήσουμε τον πίνακα αποτελεσμάτων για το δικαίωμα του καταναλωτή και διάφορα άλλα μέχρι τις 6 και 6.30 για την έκθεση του κ. Βίλαντ ε, για την γνωμοδότηση προς την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή για τον ανταγωνισμό. Καλωσορίζω την κυρία Χέντε που έχει και την σκιώδη της εισηγήτρια μαζί σήμερα την προσωπική της και Δεν έχουμε σκιώδη από το ΕΛΚ ακόμα, αλλά ελπίζω πως κάποιος θα έρθει σε λίγο. Το ΕΛΚ μπορεί να μας πει αν έχει σκιώδη, αλλά είναι αποσχολημένη η γραμματεία του ΕΛΚ συνομιλώντας. Θα έχετε κάποιον σκιώδη, θα έρθει. Ναι. Ο κύριος Μπουζό είναι εδώ, εγώ είμαι σκιώδης για τη δική μου ομάδα. Εσείς είστε, κυρία Τούρινεν, σκιώδης για τους πράσινους. Όχι, δεν έχουμε αποφασίσει. Πιθανώς, αλλά δεν έχω διοριστεί. Δεν έχετε διοριστεί. Ο κύριος Τεταφελίδης θα είναι σκιώδης για την ΚΟΕ. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Χέντ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εδώ και κάποιο καιρό έχουμε ασχοληθεί με την προστασία του καταναλωτή και να δούμε τι μπορεί να γίνει στο πλαίσιο τη Επιτροπή μα. Και την τελευταία φορά δυστυχώ ήμουν η μόνη που είχα το χρόνο να μπορέσω να εκφραστώ και περιμένω με ανυπομονησία τι παρεμβάσει του κ. Χάρμπορ αλλά και των άλλων σκιωδών εισηγητών. Θα ήθελα λοιπόν να σα πω ότι είμαι πραγματικά πολύ ικανοποιημένη που έχω αυτή τη δεύτερη εκδοχή του πίνακα επιδόσεων Έχουμε ένα ακόμα εργαλείο για να βελτιώσουμε την εσωτερική αγορά. Και τα όσα μας προτείνονται δεν είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, γιατί εδώ πρόκειται για τις προσδοκίες των καταναλωτών. Αυτό που επιθυμούν είναι να είναι πιο να λειτουργεί πιο ομαλά η εσωτερική αγορά. Κατά την άποψή μου, Υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν ώστε τα στοιχεία να είναι πιο προσβάσιμα και πιο ευανάγνωστα για τον, τον απλό αναγνώστη. Αυτό θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή προς την εσωτερική αγορά και θα το επιτρέψει και να εκμεταλλευτεί τα πλονεκτήματα. Τη τελευταία φορά σας ανέφερα τα αποτελέσματα αυτής της δεύτερης εκδοχής ε, του πίνακα, αλλά αυτό που θα πω σήμερα είναι ότι έχουμε ακριβώς στους ίδιους δείκτες με την περασμένη χρονιά όπου αυτοί χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές, η ασφάλεια σε θέματα προσφυγής και έχω ήδη πει ξεκάθαρα ότι οι καταναλωτές έχουν περισσότερο πρόβλημα με τις υπηρεσίες από ότι με τα εμπορεύματα. Πολύ συχνά υπάρχουν προβλήματα που συνδέονται με την αύξηση τιμών ή τις διασυνοριακές συναλλαγές, όπου σε ορισμένε περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε ένα ξεκάθαρο σύστημα όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων του καταναλωτή, κάτι πολύ σημαντικό για τη σωστή λειτουργία της αγοράς. Και έχω προσπαθήσει να κάνω κάποιες προτάσεις Λέω για παράδειγμα ότι θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση των οργάνων που υπάρχουν στα κράτη-μέλη σε θέματα προστασίας του καταναλωτή, γιατί στα κράτη-μέλη μας υπάρχουν πραγματικά μεγάλες διαφορές όσον αφορά τις δομές που είναι στη διάθεση των καταναλωτών και ελπίζω πως τα όσα προτείνω θα επιτρέψει να αυξηθεί η διαφάνεια και θα μας δείξει τι είναι πραγματικά απαραίτητο για να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Από τη στιγμή που έχουμε ισχυρούς καταναλωτές είναι δυνατόν να παρακολουθήσει κανείς τις διασυνοριακές συναλλαγές και πιστεύω πως από την άποψη την νομική θα πρέπει επίσης να βρούμε εναλλακτικέ στις, ε, ε, στις περιπτώσεις ε, αντιπαράθεσης. Δεν θα πρέπει πάντοτε να καταφεύγει κανείς στα δικαστήρια όταν πρόκειται για κάποιο πρόβλημα και ακόμα περισσότερο τώρα που διανύουμε κρίση η κατάσταση του καταναλωτή είναι πολύ πιο ευάλωτη από ό,τι συνήθω. Έχουμε πολλούς καταναλωτές που εμπλέκονται εδώ σε δίκες, πράγμα που τους κοστίζει χρόνο και χρήμα και θα έπρεπε να μπορούμε να βρούμε μια εναλλακτική λύση για τον καταναλωτή αλλά και για τις εταιρείε. Επίσης νομίζω θα πρέπει να συζητήσουμε το CPS. Αυτή τη φάση δεν έχω συγκεκριμένε προτάσει να σας κάνω, αλλά έχω την εντύπωση πως θα πρέπει πραγματικά να ακολουθήσουμε την πορεία μιας ε, αυξημένης συνεργασίας. Τελευταία μου παρατήρηση να πιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι αυτός ο πίνακας δεν χρηματοδοτείται πραγματικά όπως το κάναμε και στο πλαίσιο της τελευταίας μας σύστασης και θα πρέπει να γίνει μια έκκληση προς τα κράτη-μέλη ώστε να μεριμνήσουν για να υπάρξει κατάλληλη χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και σε εθνικό επίπεδο γιατί χωρίς έλεγχο της αγοράς η κατάσταση μπορεί να είναι αρνητική για τον καταναλωτή και αν θέλουμε η εσωτερική αγορά να λειτουργήσει θα πρέπει να έχει ο καταναλωτής εμπιστοσύνη σε αυτή την αγορά. Χωρίς κάτι τέτοιο δεν θα έχουμε νυφάλους καταναλωτές. Και να πιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι την περασμένη φορά όταν υιοθετήσατε τα αποτελέσματα του πίνακα αποτελεσμάτων δεν υπήρχε πρόβλημα και πιστεύω πως τα αποτελέσματα είναι πραγματικά εξαιρετικά. Έχουμε μια νέα επιτροπή που σε λίγο θα είναι εδώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιμείνουμε για τη σημασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Δεν θα πρέπει το σημείο αυτό να εξαφανιστεί στο μέσο άλλων θεμάτων που θα θυγούν από πλευρά της Κομισιόν. Αυτά είχα να σας πω κύριε Πρόεδρε και περιμένω να ακούσω και τις ε, παρεμβάσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ που συνεχίζετε τη δουλειά που ξεκινήσατε πριν από μερικές εβδομάδες. Ο κύριος Μότι είναι εδώ. Ο κυρία Τούρινεν και εγώ και ο κύριος Τριανταφυλλίδης είμαστε σκιώδης. Να καλωσορίσω και τον David May από πλευρά τη Κομισιόν που πιστεύω ότι θα είναι ο βασικός μας συνομιλητής από πλευρά της Κομισιόν γιατί είναι ο αρχιτέκτονας αυτού του πίνακα αποτελεσμάτων καθώς συζητάμε και την ανακοίνωση για την επιβολή επίσης. Θέλετε να μιλήσετε λοιπόν για όλα αυτά, θα είστε ευπρόσδεκτος. Κύριε Μότι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά σύντομος γιατί θεωρώ πως ε, το κλίμα εντό του οποίο αντιμετωπίζουμε αυτό το, την έκθεση μπορεί να είναι πλήρως συνεργασίας και διαλόγου γιατί Νομίζω πως θα πρέπει όλοι να συμφωνούμε για το γεγονός ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να τους δίνεται ε, μια μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής να προστατεύονται από κάθε πλευρά και εδώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να είμαστε πάντοτε προσεκτικοί, να μην τους επηρεάσουμε, δηλαδή να μην τους υποκαταστήσουμε στην ε, απόφασή τους και παράλληλα να εγγυηθούμε τις ε, προϋποθέσεις για μια ελεύθερη αγορά που επιτρέπει στους ανταγωνιστές να προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα με το μικρότερο δυνατό κόστος, γιατί και αυτός είναι ένας τρόπος για να αυξηθεί η ελευθερία των καταναλωτών και για να προστατευθούν. Επίσης πιστεύω πως ε, πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε μια προσέγγιση εναρμόνισης ε, με τους όρους που θα εντοπίζουμε, γιατί είναι σαφές ότι κάθε κράτος θα προσπαθήσει να λύσει τα εσωτερικά του προβλήματα, αλλά εμείς ε, ασχολούμαστε με τους Ευρωπαίους καταναλωτές και από αυτή την άποψη είδα να υπάρχει κάποιος περιορισμός, που είναι περιορισμός της βάσης δεδομένων, περιοριστική βάση δεδομένων που έχει ληφθεί υπόψη, για να δουλέψουμε πάνω σε αυτή την έκθεση είδα ότι δεν υπάρχει μια πλήρη ομοιογένεια και αυτό σίγουρα αποτελεί έναν περιορισμό γιατί εμείς θέλουμε να κάνουμε πλήρη εργασία και δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε στοιχεία τα οποία είναι σχετικώς ε, ατελή ή επί των που δεν είναι συγκρίσιμα. Ε, και από αυτή την άποψη λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε πως θα χρειαστούν παραπάνω πόροι ακριβώ για να διευρυνθούν τα κριτήρια συλλογής αυτών των στοιχείων επί των οποίων εμείς θα βασίσουμε τη δικιά μας δουλειά γιατί σίγουρα χρειάζεται ομοιογένεια για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια για το ποιοι θα είναι οι στόχοι μας. Φυσικά ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε και καλύτερη δουλειά αν μπορούσαμε να ευνοήσουμε μια ανταλλαγή πληροφοριών για την αριστεία, γιατί θα πρέπει να έχουμε υπόψη πως οι καταναλωτές ε, λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι για ορισμένα προϊόντα και κυρίως για τις ε, τραπεζικές υπηρεσίες, τραπεζικές, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις μεταφορές κτλ. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν πάνε όλα χάλια, όπου υπάρχει αριστεία ακόμα και σε κάποιους τέτοιους μεμονωμένους τομείς. Το να δουλέψουμε σωστά θα σημαίνει ότι θα θέσουμε στη διάθεση των καταναλωτών όλων των χωρών της Ένωσης τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την εμπειρία που τη θετική στις χώρες όπου οι τομείς αυτοί δεν πήραν αρνητικό βαθμό. Μεγαλύτερη συνεργασία σίγουρα και μεταξύ των κρατών μελών από αυτή την άποψη και συντονισμός ανάμεσα που είναι μάλλον απαραίτητος ανάμεσα στην Κομισιόν και το Κοινοβούλιο και με τους ε, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμενες για να κάνουμε μια πραγματική ε, συμβολή. Θα πρέπει επίσης να αναλύσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο γιατί και εκεί οι καταναλωτές δεν έχουν αρκετή εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει αρκετή προστασία. Και θα χρειαστεί να εργαστούμε για να αγγιηθούμε την ε, βοήθεια μετά την πώληση, γιατί ένα πρόβλημα που έχει καταγγελθεί είναι το πρόβλημα της έλλειψης ε, απάντησης όταν γίνεται κάποια καταγγελία ή αμφισβήτηση από πλευρά του καταναλωτή. Δηλαδή δεν είναι θέμα μόνο τη παροχή τη υπηρεσία, αλλά και το πώ ε, δίνεται συνέχεια η απάντηση στην ανάγκη του, του, καταναλωτή που θεωρεί που δεν έχει εξυπηρετηθεί σωστά. Παραλαμβάνω, σε ένα κλίμα συνεργασία και διαλόγου θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε ποιε είναι ανάγκε για να εγγυηθούμε στου καταναλωτέ αλλά και στου προμηθευτέ των υπηρεσιών και στου παραγωγού, ε, έτσι ώστε να δίνεται σε μια απόλυτα ελεύθερη αγορά η καλύτερη δυνατή υπηρεσία προς τον καταναλωτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη του κυρίου Ροσφόρ, ο οποίος είναι ο σκιώδης μας ε, και για αυτή την έκθεση και για την έκθεση ΣΒΑΜ, διότι απουσιάζει αλλά υπάρχει μια πολύ σημαντική ε, τελετή στη χώρα του και δεν μπόρεσε να έρθει. Θα ήθελα τώρα να, να κάνω όμως μερικά σχόλια. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το δεύτερο πίνακα βαθμολόγησης και ε, να πω ότι είναι πολύ βασικός ε, και για τους πολιτικούς, για τους διάφορους, ε, για τις διάφορες τάξεις και για τους καταναλωτές που έχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να υπάρχει μία γενική επισκόπηση του και ένας πίνακας βαθμολόγησης σχετικά με την προστασία των καταναλωτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι εδώ μιλάμε για υποκειμενικές συμπεριφορές, έχουμε διαφορετικές συμπεριφορές στα διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ίσως όταν θα υπάρχει μία ενιαία νομοθεσία και υιοθετηθεί η οδηγία θα ε, είναι πολύ πιο σημαντικό το θέμα αυτό αλλά ε, εάν θέλουμε να κοιτάξουμε τουλάχιστον τους δείκτες των παραπώνων και της ικανοποίησης πιστεύω ότι είναι πολύ ε, υποκειμενική. Κοίταξα λοιπόν στη Ρουμανία, στη χώρα μου δηλαδή και βλέπω ότι εκεί υπάρχουν ε, λιγότερα παράπονα από ότι μικρότερες χώρες. Διότι όπως σας είπα Έχουμε διαφορετική αξιολόγηση, διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικό τρόπο αξιολογήσεως και όλοι οι πολίτες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και δεν ε, θέλουν όλοι οι Ευρωπαίοι ε, πολίτες να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους ε, σε όλες τις χώρες το ίδιο. Όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο, παρόλο που ακόμη 57% των ε, Ευρωπαίων καταναλωτών λένε ότι δεν ενδιαφέρονται ε, να κάνουν μια διασυνοριακή αγορά τους επόμενους 12 μήνες. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο εφέτος και κάθε χρόνο όλο και περισσότερο οι καταναλωτές ε, δεν έχουν αντίρρηση να ψωνίζουν διασυνοριακά και γι' αυτό υπάρχει ένας ε, σοβαρός λόγος για την εσωτερική αγορά να εκδώσει αυτή την νομοθεσία κατά τρόπον ώστε να ξέρουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, τα βασικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Κατά τα άλλα όμως πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και είμαι βέβαιος ότι θα μας δοθούν και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Η κυρία Τούριν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. είναι λιγάκι έκπληξη ότι ε, μου ζητήσα τώρα το λόγο. Δεν έχω τόσα πολλά να πω. Στηρίζουμε βεβαίως την δουλειά της εισηγήτριας. Τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά. Η πληροφόρηση και πρέπει να δούμε τι χρειάζεται στην νομοθεσία, να το επεξεργαστούμε ή τι νέα ενάυσματα πρέπει να προσφέρουμε. Ε, ερχόμαστε τώρα στη χρηματοδότηση, η οποία εξαρτάται από τα κράτη-μέλη. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και γι' αυτό χρειαζόμαστε και την ε, ε, χρηματοδότηση και από ό,τι κατάλαβα ορισμένοι δείκτες είναι πολύ υποκειμενικοί. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε τους ποιοτικού παράγοντες διότι το θέμα είναι πώς αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τα μέτρα αυτά και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο να μετρηθεί. Υπάρχει και διαφορετικό σημείο κινήσεως αναλόγως του κράτους. Ε, πρέπει να είμαστε εδώ φιλόδοξοι, να κοιτάξουμε να βελτιώσουμε ό,τι έχουμε ήδη και να διατυπώσουμε φιλόδοξες προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τούριν που αναλάβατε αυτή την ευθύνη. Ξέρω ότι η κυρία Ρούλε είναι η σκιώδηση για πάρα πολλά θέματα και γι' αυτό ε, ε, χαίρομαι που θελήσατε να ε, επέμβετε. Ε, τώρα εγώ θα ήθελα να πω ότι κατόπιν της εξελίξεως προηγούμενο, στην προηγούμενη θητεία του Ευρωκοινοβουλίου είχα ορισμένες επιφυλάξεις για αυτό το θέμα. Αλλά τώρα φτάνουμε σε κάποιο σημείο όπου όντως θα αποτελέσει ένα πολύ βασικό στοιχείο πολιτικής και αυτή η εργασία ουσιαστικά επικεντρώνεται στα ιστορικά στοιχεία. Δηλαδή διαπιστώνουμε δείκτες ε, για αλλαγές και αν, ακόμη και αν δεν είναι ουσιαστικές αλλαγές, ορισμένες αλλαγές έχουν ήδη εντοπιστεί και από πλευράς πληροφόρησης θα είναι πολύ βασικό να μπορούμε να παρακολουθούμε την πληροφόρηση. Θα είναι δηλαδή βασικό να διατηρήσουμε την ε, ουσία ε, του θέματος σταθερή προς το παρόν και θα δούμε που θα μας βγάλει θα δούμε στις, ε, εάν στις δύο ή τρεις επόμενες μετρήσεις οι δείκτες δεν ε, μας χρησιμεύουν, μήπως θα, θα χρειαστεί να τους αξιολογήσουμε και να τους αλλάξουμε. Και οι τιμές ε, είναι σημαντικές. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ορισμένα στοιχεία της έρευνας του καταναλωτούν όσον αφορά την αντίληψη ε, των κυβερνήσεων για το θέμα ε, διαφέρει πάρα πολύ και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές αντιμετωπίσεις των καταναλωτών αναλόγως των χωρών. Λοιπόν, η μορφή αυτού του είδους ε, της εκθέσεως είναι πολύ χρήσιμη. Είναι βασικό να έχουμε ουσιαστικά στοιχεία και κάθε χρονιά να προχωράμε περισσότερο εις βάθος. Ε, κάθε χρόνο δηλαδή θα πρέπει να συνδυάζουμε τις μετρήσεις αυτές με μία συγκεκριμένη ειδική μέτρηση. Θα πρέπει δηλαδή να εξετάσουμε ορισμένα στοιχεία, ε, παραδείγματο χάρη, γιατί ορισμένοι καταναλωτές σε ορισμένες χώρες θεωρούν ότι είναι πιο προστατευμένοι από ό,τι αλλού. Γνωρίζουν καλύτερα τα δικαιώματά τους έχουν κάποιον στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν, ένα διαμεσολαβητή, ε, κάποιον ε, εξέχοντα. Υπάρχει μία πολύ ισχυρή οργάνωση καταναλωτών στη χώρα αυτή νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό να ε, συσχετίσουμε όλα αυτά τα στοιχεία γιατί αυτό θα ενδιαφέρει την Επιτροπή ε, φαντάζομαι γιατί έτσι θα ξέρουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη δραστηριότητά μας και πώς θα εμπλακούμε περισσότερο για να ικανοποιήσουμε τους καταναλωτές. Όσον αφορά τα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα για τις υπηρεσίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες, νομίζω ότι είναι ένα θέμα πολύ χρήσιμο διότι άπτεται και των ευθυνών της δικιάς μας Επιτροπής που αναφέρεται εις ε, τις προδιαγραφές ποιότητος και πρέπει να ενθαρρύνουμε ε, τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν προδιαγραφές ποιοτικέ για τις υπηρεσίες. Από άλλα στοιχεία βλέπουμε κατά πόσον η ε, ικανοποίηση του καταναλωτή συνδυάζεται με την ε, ανυπαρξία στοιχείων ή την ανεπάρκεια των στοιχείων μπορεί σε ορισμένα πράγματα ε, να υπάρχουν έννοιες οι οποίες είναι άειλες αλλά σε ένα προϊόν παραδείγματο χάρη μπορείτε ενδεχομένω να το δοκιμάσετε πριν το αγοράσετε. Εάν αγοράσετε ένα κινητό τηλέφωνο π.χ. έχετε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο γενικά και ε, γενικότερα και αυτό είναι ένα διαφορετικό ερώτημα που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι προφανές ότι είναι πολύ χρήσιμο αυτό το στοιχείο για τους ε, νομοθέτες. Και ίσως υπάρχουν πτυχές οι οποίες ακόμη δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς. Αυτό που είναι βασικό για μας είναι, ε, υπάρχει ένα πιο δημοφιλές μήνυμα το οποίο μπορεί να διατυπωθεί και ποιος είναι ο στόχος ε, πρέπει να είναι ε, ένα ευρετήριο για τους για τους ηθήνοντες και τους νομοθέτες για να μπορέσουν να το συμβουλεύονται ή για το Κοινοβούλιο μπορεί να είναι ένας χρήσιμος δείκτης για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν καλύτερα με τους καταναλωτές και να τους ενημερώσουν. Δηλαδή νομίζω ότι ορισμένα από τα θέματα εδώ είναι γενικότερα και καλό θα ήταν αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να απευθυνθεί εις το ακροατήριο και να διερευνήσει αν χρειάζεται μία πιο ε, λαϊκή μορφή της εκθέσεως. Επίσης, όπως είπα προηγουμένως, ε, είναι, εύκολο να δούμε πόσο ορισμένοι ε, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διορθωτικές κινήσεις και σε αποκατάσταση ε, κάποιας ε, ζημίας και νομίζω ότι τώρα η συγγήτρια που έχει το δύσκολο έργο να συνδυάσει όλες τις πτυχές ε, θα έπρεπε να μας ε, ενημερώσει από αυτόν. Εχθές όμως αναφέρθηκα στο δίκτυο για την συνεργασία των καταναλωτών που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες και κατάρτισε το πρόγραμμα συνεργασίας για την περίοδο 2009-2010 και τους διαβεβαίωσε για το πόσο σοβαρά εξετάζεται σε αυτή την Επιτροπή αυτό το θέμα, ιδίως διότι η ουσιαστική νομοθεσία που οδήγησε σε αυτή την οδηγία ήταν το πρόγραμμα της κυρίας Γκέμπχαρτ, το οποίο παρακολούθησε προσωπικά. Είπα επίσης ότι έγινε μία παρουσίαση ε, και λάβαμε ένα αντίγραφο αυτής της έκθεσης προσφάτων, προσφάτως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει να σκεφτεί μακροπρόθεσμα τη στρατηγική της και ίσως εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τι άλλα πράγματα μπορούμε να ε, κάνουμε από αυτού. Δηλαδή ε, μιλήσαμε και στο παρελθόν ε, για διάφορα θέματα, ε, για ε, διευκρινήσεις, sweeps, που είναι ένας τρόπος να εξηγήσουμε κάτι και να το καταλάβουν οι καταναλωτές θα πρέπει να συνδυάσουμε τις ενέργειες αυτές ε, με στρατηγικές ενέργειες που θα προσεγγίσουν το καταναλωτή πιο αποτελεσματικά από ό,τι τώρα και θα συνδυαστούν με τη διάθεση μεγαλύτερων οικονομικών πόρων. Ε, το ίδιο που είπαμε και το πρωί για το Solvit για να μπορέσουν να μας ε, ε, συνδράμουν οι κυβερνήσεις και για να μπορέσουμε να αναφερθούμε σε περισσότερα θέματα. Εδώ νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την καλή της δουλειά. Αυτά είχα να πω σαν εισηγητής και τώρα παρακαλώ τον κύριο Τριανταφυλλίδη εν ονόματι της ΓΚΟΕ να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σε αυτό το αρχικό στάδιο της ανταλλαγής απόψεων θα περιοριστώ να πω ότι η προστασία των καταναλωτών είναι για τη δική μας ομάδα ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Να υπενθυμίσω ότι ως ομάδα κάναμε μια πρόταση για έναν initiative για τον έλεγχο των τιμών, κάτι που βασικά κάνει ο πίνακας αυτός οπωσδήποτε θα συνεργαστούμε πλήρως με την ε, εισηγήτρια για να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε, αν μπορώ να πω έτσι, την ε, εργασία για να πούμε και εμείς τις δικές μας απόψεις που ελπίζω να σωματωθούν τελικά στο κείμενο. Ε, ο πίνακας φαίνεται να είναι ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν πολιτικές προεκτάσεις από την ερμηνεία που μπορούν να έχουν τα αποτελέσματα για τις τιμές. Ε, θα συμφωνήσω με ένα σημείο που έγινε προηγουμένως ότι δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να καθοδηγήσουμε τον, τις επιλογές του καταναλωτή αν και ο πίνακας θα πρέπει να είναι ενδεικτικός των αποτελεσμάτων και να παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσματα. Επομένως, ως ε, πολιτική ομάδα θα παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά τις μεταβολές των ε, τιμών και θα πρέπει να ενδυναμώσουμε αυτό το εργαλείο που μας προσφέρει ο πίνακας για την προστασία των καταναλωτών. Ευχαριστώ πολύ. Well, θέλουν να παρέμβουν άλλα μέλη. Εάν ε, όχι, ίσως ο κύριος Μέρ θα πρέπει να σχολιάσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρου σας που σας είπατε ότι εγώ ήμουν αρχιτέκτονας του scoreboard. Νομίζω όμως ότι η πραγματική αρχιτέκτον ήταν η Επίτροπος κυρία Κουνέβα. Ε, ήταν δική της ιδέα και από εκείνη ξεκίνησε αυτό το έργο. Και νομίζω ότι σωστάμε πολλά για αυτή την ε, ε, κατανόηση που είχε όσον αφορά την πρόθεση των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση ακριβώς με τη συλλογή αυτών των δεδομένων που αναλύουν τη θέση των καταναλωτών στις αγορές. Και η δημιουργία αυτών των δεδομένων θα είναι η κινητήρια δύναμη και ο γνώμονας βάση του οποίου θα δούμε κατά πόσο έχουν γίνει κατανοητά, κατανοητές οι ανάγκες των καταναλωτών. Νομίζω ότι πραγματικά τις χρωστάμε πάρα πολλά για αυτή την ε, ιδέα. Η, υπό την έννοια αυτή η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου έρχεται πραγματικά ε, στη σωστή ώρα και είναι σαφές από τις κατευθυντήριες γραμμές ότι το θέμα της ε, παρακολούθησης της αγοράς και ο ρόλος του πολίτου ε, θα βρίσκονται στο επίκεντρο των προβληματισμών του επόμενου επιτρόπου σε σχέση με, ε, το πρόγραμμα 22 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την έκθεση Μόντι. Εάν θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε τη θέση των καταναλωτών η παραγωγή μιας, ε, η δημιουργία μιας ε, καλά τεκμηριωμένης ε, ανάλυσης θα μας αποδεικνύει κατά πόσο λαμβάνονται παρκώς υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών, τα οποία δεν είναι μια λεπτομέρεια. όταν εξετάζουμε θέματα ανταγωνισμού, εσωτερικής αγοράς, καινοτομίας ή ολοκλήρωσης ακόμα, η διάσταση του καταναλωτού είναι εξαιρετικά σημαντική σε σχέση με όλα αυτά και θα πρέπει να συλλέξουμε σωστά τα δεδομένα ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την σωστή κατανόηση της θέσης των καταναλωτών. Ε, η δεύτερη έκδοση του πίνακα κινείται απλώς στην επιφάνεια ε, και νομίζω ότι ε, μελλοντικά θα μπορέσουμε να φτιάξουμε το είδος του πίνακα το οποίο όλοι αναμένουμε. Ε, ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι, έχει κατέχει μια θέση κλειδί. Ε, θέλουμε να έχουμε δεδομένα τα οποία να είναι καθοριστικά σε εθνικό αλλά και, και ωφέλιμα σε εθνικό αλλά και σε κοινοτικό επίπεδο. Θα ήθελα τώρα να σα δώσω μια πρόγευση για των σημαντικών προγραμμάτων τα οποία θα εκπονήσουμε τι προσεχεί ε, μήνες. Καταρχήν σε σχέση με τις τιμές. Τώρα ξεκινούμε να διαπιστώνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα απέχει πάρα πολύ από την ε, δυνατότητα να παραγάγει ένα αξιόπιστο σύστημα τιμών. Προσπαθούμε λοιπόν να να, να εκπονούμε κάποιους ε, δείκτες. Νομίζω ότι προσεχώς θα δούμε στην επόμενη επιτροπή την έγκριση μιας ε, σύστασης που θα περιλαμβάνει όλα τα σώματα ε, διαχείρισης των παραπώνων εκ μέρους των καταναλωτών. Ε, υπάρχει μια πληθώρα αυτών των παραπώνων που συλλέγονται με διάφορους ε, τρόπους. Ε, προσπαθούμε να δουλέψουμε στη βάση μιας εναρμονισμένης μεθοδολογίας που θεωρούμε ότι θα είναι ιδιαίτερως χρήσιμη και ελπίζουμε ότι τον επόμενο χρόνο θα μπορέσουμε να έχουμε επίκαιρα, ε, ε, επικαιροποιημένα δεδομένα που θα μας ενημερώνουν επαρκώς για τις καταγγελίες και τα παράπονα των Ευρωπαίων πολιτών εκεί όπου πραγματικά ε, χρειάζεται μια παρέμβαση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όσον αφορά την πρόσληψη των καταναλωτών σε σχέση με τις προβληματικές αγορές, η Δανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Σουηδία, εσείς που προέρχεστε από αυτές τις χώρες, ε, θα γνωρίζετε ε, το θέμα αυτό που δίνει δυνατότητα ε, στους πολιτικά ηθήνοντες να αναγνωρίζουν τις προβληματικές αγορές. Κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν κάποιες επιλογές. Ε, από τον επόμενο χρόνο θα υπάρχει μια ιεράρχηση των 15 αγορών, 15 ε, αγορών και θα είναι διακριτή η θέση της κάθε χώρας, ε, βάσει της οποίας θα εντοπίζονται τα επακριβώς τα προβλήματα της εσωτερικής αγοράς. Τώρα, δύο άλλα θέματα. Η Eurostat εκπονεί μία μελέτη η οποία εξετάζει τις δεξιότητες ε, των καταναλωτών και τις δυνατότητες ενίσχυση των καταναλωτών. Κατά πόσο οι καταναλωτές γνωρίζουν τις δυνατότητές τους, ε, ε, γνωρίζουν ότι μπορούν να επιστρέψουν κάποια είδη, είναι παρκώς ενημερωμένοι. Αυτή η έρευνα θα γίνει τους, τους πρώτους τρεις μήνες του 2010 και θα μας ενημερώσει για τα προβλήματα των καταναλωτών που ακριβώς θα πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειες χώρες μέλη για να εκπαιδεύσουν, να καταρτήσουν τους καταναλωτές. Κατά δεύτερο λόγο, ξεκινά μια πιλωτική έρευνα της αγοράς, ο σκοπός του scoreboard ήταν να μας δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και να ανοιχνεύσουμε τους ε, τομείς που παρουσιάζουν προβλήματα. Αλλά αυτή τη στιγμή γίνει αυτό, μπορούμε να πάμε εις βάθος και να μελετήσουμε πού ακριβώς εντοπίζονται το προβλήματα των καταναλωτών. Ε, καταρχήν θα ξεκινήσουμε από την αγορά του ηλεκτρισμού και ε, της ηλεκτρικής ενέργειας και ελπίζουμε μέχρι το φθινόπωρο να είναι εγκλωγρωμένη αυτή η έρευνα και να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε παρκώς τα προβλήματα των καταναλωτών σε σχέση με την, παροχή, με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ούτω ώστε να μπορέσουμε να αντιδράσουμε με ταχύτητα στα προβλήματα αυτά και να μπορούμε να αναγνωρίζουμε με επιτόπιους ελέγχους τα προβλήματα ει βάθο. Τέλος, ε, θα ε, χρειαζόμαστε βεβαίως περισσότερη ανάλυση σε σχέση με τα δεδομένα αυτά. Ένα από τα συμπεράσματα στο οποία καταλήξαμε είναι ότι έχουμε μια πληθώρα πληροφοριών που περιέχονται στο πίνακα, στο scoreboard και αυτό το οποίο αποφάσισε η Επίτροπος Κουνέβα είναι να προσεχώς το scoreboard να βγαίνει σε δύο τμήματα. Το πρώτο, το Μάρτιο του προσεχούς έτους που να εστιάζει ε, σε προβλήματα που αναφέρθηκαν στη ΣΥΤΣΙ, δηλαδή πού εντοπίζουν ακριβώς τα προβλήματα στο επίπεδο των χωρών μελών. Ε, το παρόν ε, τμήμα 2 και 3 του scoreboard. Μία ενημέρωση εν σχέση που βρισκόμαστε στον αφορά του διασυνορικό εμπόριο, αλλά επίση θα εξετάζει την απόδοση, την αποδοτικότητα μάλλον των εθνικών οργανισμών και επίσης θα πηγαίνει πίσω από πράγματα που αναφέρετε εσείς κύριε Πρόεδρε, δηλαδή ε, πού ακριβώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ε, στις συγκεκριμένε. χώρες. Και αργότερα τον Οκτώβριο θα έχουμε το scoreboard το οποίο θα κάνει μια εράρχηση των αγορών ε, σε συνάρτηση με, τα, με την αναγνώριση των προβλημάτων για τους καταναλωτές. Και στη βάση αυτή μπορούμε να επιλέξουμε έναν τομέα όπου χρειάζεται μια περισσότερη βάθος μελέτη. Εν συντομία, ο δεύτερο, το δεύτερο scoreboard είναι καρπός 12 μήνες εργασίας αυτής της ομάδας. Ο επόμενος πίναξ, ο επόμενο scoreboard ε, θα έχει ευρύτερο φάσμα δεδομένων. Ε, ελπίζω θα μπορέσουμε να τηρήσουμε τις προθεσμίες. Ε, προφανώς χρειάζεται μια ε, παρακολούθηση αυτών των δικτών, να δούμε πώς εξελίσσονται και ελπίζουμε ότι μελλοντικά θα έχουμε με περισσότερες βάθους ανάλυση η οποία θα είναι πιο κοντά στην διατύπωση ε, πολιτικών συστάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και την ε, Επιτροπή σας, ε, και την, καθώς και σας κύριε Πρόεδρε για την, ε, το προσωπικό σας ζήλο. νομίζω ότι η συζήτηση αυτή για τον προγραμματισμό του επόμενου έτους και ακόμα παραπέρα είναι ιδιαίτερος χρήσιμη. Ήταν πολύ χρήσιμη η επίσκεψη μας εδώ. και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί και τη δική μας εργασία και τον τρόπο που την επιτελούμε. Η ανακοίνωση για την εφαρμογή επισημαίνει τα πιο σημαντικά ε, ευρήματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων. Όπως είπε η κυρία Κούνεβα, ε, ο νόμος βρίσκεται στα καρτιά. Ε, δεν θα έχει μεγάλη σημασία για τον καταναλωτή χωρίς την εξουσία ε, για την εκτέλεσή του, την εφαρμογή του. Η παρούσα κρίση δίνει ένα πολύ καλό παράδειγμα για το όσον αφορά ε, το θέμα της ε, εκτέλεσης. αν η εκτέλεση γίνεται μόνο η εφαρμογή σε περίοδους κρίσης, τότε είναι αναποτελεσματική. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα τα οποία εκχωρούνται πράγματι να εκπληρώνουν, να πληρούνται, να εφαρμόζονται, ούτως ώστε να υποφελούνται όλοι. Όπως επισημάνθηκε ήδη η εφαρμογή εναπόκειται στην ευθύνη των χωρών μελών κατ' ουσία. Στον τομέα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού αλλά ε, λειτουργούν, αλλά μόνο ε, τα δύο όργανα δεν μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα. Θεωρώ ε, ότι είναι πολύ σημαντική δική συμμετοχή στο, στη διαδικασία αυτή και είμαι ευγνώμων που θεωρείται, όπως αναφέρθηκε σήμερα το απόγευμα, ότι θα συμμετάσχετε στην αξιολόγηση του προγράμματος και εγώ από την πλευρά της Επιτροπής είμαστε στη διάθεση να συνδράμουμε σε αυτή τη διαδικασία. Μια και αναφέρεται το ζήτημα του προγραμματισμού, ε, πράγματι βρίσκεται υπό εξέλιξη. Ε, κάναμε ένα σχέδιο εφαρμογή για το επόμενο έτος, χθες το αποφασίσαμε και συμφωνήσαμε για λόγους ασφάλειας. Δεν θα ήθελα τώρα να σας ανακοινώσω το θέμα, αλλά θα είναι πολύ ενδιαφέρον, μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Τώρα, όσον αφορά τα ζητήματα εφαρμογής, ε, επιτεύθηκε συμφωνία και σε άλλα θέματα αφορούν την προστασία των καταναλωτών. Συμφωνήσαμε να έχουμε κοινέ ε, δράσεις όπου οι συνθήκες ε, μπορούν να ε, ε, οδηγήσουν στην έναρξη μιας διαδικασίας. Επίσης, συμφωνήσαμε με την οργάνωση ορισμένων workshops σε σχέση με την εφαρμογή διαφόρων ευρωπαϊκών συστημάτων δικαίου, καθώς και για ζητήματα προστασίας καταναλωτών σε σχέση με τα λεγόμενα green claims. Επίσης, ε, ε, αποφασίσαμε να συστήσουμε δύο ομάδες εργασίας για διαφορετικά θέματα, ούτως ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τι ακριβώς σημαίνει και να μπορέσουμε να απευθύνουμε κάποιες προτάσεις προς τους νομοθέτες. Ε, χθες ήταν μια πολύ γόνιμη ημέρα, μπορώ να σας πω, και τον επόμενο χρόνο θα έχουμε θετικά αποτελέσματα, ελπίζω, και θα μπορέσω να σας τα ανακοινώσω προσεχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θετικά σας σχόλια. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και πιστεύω ότι δείχνω ότι η Επιτροπή από κοινού με τις χώρες μέλη βρίσκονται στο σωστό δρόμο και ελπίζω το πρόγραμμα για το επόμενο έτος και ακόμα παραπέρα θα συμβάλλουν στη βελτίωση του επίπεδου προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα... Να σας ευχαριστήσω για τις ε, πολύ τομένες σας απαντήσεις και για τις φρέσκες σας ιδέες. Λοιπόν, θα θέλατε τώρα να ολοκληρώσετε. Έχουμε λίγο χρόνο στη διαθεσή μας. Αν θέλει κάποιος άλλος το λόγο, να σας δώσω το, το λόγο. Όχι. Αν θέλετε λοιπόν να συνοψίσετε και να μιλήσουμε και για το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί η κόρη μου και εγώ Είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε το αεροπλάνο για τη Σουηδία σε λίγες ώρες και πιστεύω όπως το είπατε και όπως το είπε και η Κομισιόν πολύ σωστά, αυτό που είναι σημαντικό είναι να γνωρίζουμε το γεγονός ότι τα όσα έχουμε εδώ είναι ένα νεογέννητο, ένα μωρό Όταν θα μεγαλώσει θα είναι πολύ σημαντικό, θα βοηθήσει πολύ για την ε, εσωτερική αγορά και θα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι είμαστε στις αρχές των εργασιών. Και ε, όπως είπατε είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετική στάση. Όταν πρόκειται για την έννοια της του, της προστασίας ε, του καταναλωτή θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε μια σχετική μελέτη. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο των εργασιών μας να δούμε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μπορέσουμε και να συνεργαστούμε με ΜΚΟ και με οργανισμούς που ήδη γνωρίζουν πολλά πράγματα. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε αυτή τη σημαντική συζήτηση θα πρέπει να συνεργαστούμε με άλλους εταίρους. Για το χρονοδιάγραμμα δεν το έχω να μου. Προσπαθώ να συντάξω ένα κείμενο που θα πρέπει να είναι έτοιμο για να σταλεί στην μετάφραση τον Ιανουάριο. Αλλά αν έχετε συγκεκριμένες ημερομηνίε να μας διαβιβάσετε, φυσικά μπορείτε να μας τις πείτε και να μας τις θυμίσετε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Νομίζω πως συμφωνούν οι προτινόμενες ημερομηνίε. Ελπίζω πως θα μπορείτε να ε, μας στείλετε την έκθεσή σας για μετάφραση μέχρι τις 7 Ιανουαρίου να το εξετάσουμε στη συνεδρίασή μας ανάμεσα στις 25 και 26 Ιανουαρίου. Είπαμε ότι μπορεί να υπάρξει και μια ειδική ε, συνεδρίαση για να εγκρίνουμε την Επιτροπή. Εάν βέβαια υποθέσουμε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ακροάσεις και ότι το Κοινοβούλιο θα έχει λάβει τις ε, ε, αποφάσεις του κτλ. Θα το δούμε, μας περιπτώσει τη τελευταία στιγμή. Και να περάσει από την Ολομέλεια το Μάρτιο. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο χρονοδιάγραμμα και για το σχεδιασμό της έκθεσης για την ε, συνεργασία των καταναλωτών. Η έκθεση αυτή μπορεί να είναι ακόμα μία μέθοδος για να έχουμε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το ποιοι είναι οι στόχοι και οι φιλοδοξίες για τα διάφορα στοιχεία της πολιτικής προστασίας του καταναλωτή εντός της Κομισιόν. Αυτά βέβαια είναι θέματα που θα τα εξετάσει ο νέος Επίτροπος. Συμφωνείτε με το χρονοδιάγραμμα. Ωραία. Θα σας στείλω και τα στοιχεία αυτά και οι σκιώδεις φυσικά θα συναντηθούν μαζί σας για να τα συζητήσετε όλα αυτά πριν ε, συνεχιστεί η εργασία σας. Ε, τώρα, ο Άντρος Βάμπ είναι εδώ. Θα δώσω την προεδρία στην κυρία Βερνιό Μήπως μπορείτε να μας δώσετε δύο λεπτά για να αλλάξουμε θέση εδώ στο Προεδρείο. Θα ξεκινήσουμε στις 4. με την έκθεση για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Λοιπόν, τελειώνει το σύντομο διάλειμμα το οποίο κάναμε, γιατί θα ασχοληθούμε με ένα θέμα πολύ σημαντικό. Έχουμε χρόνο για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε σωστά. Είναι ο φάκελος των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Έχουμε δύο ώρες για να το συζητήσουμε. Δηλαδή θα είμαστε πολύ λιγότερο περιορισμένοι από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις. Κύριε Σβάμπ, είσαστε λοιπόν ο εισηγητής για τα δικαιώματα των καταναλωτών, ένα πολύ βασικό θέμα για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και πιστεύω ότι σήμερα εσείς προτείνατε να εστιάσουμε τη συζήτησή μας και αυτό είναι πολύ ουσιαστικό στο κεφάλαιο 4 αυτής της οδηγίας η οποία ονομάζεται άλλα δικαιώματα των καταναλωτών που αναφέρονται εις ε, ε, το συμβόλαιο πολίσεως. Είναι συγκεκριμένο, οπότε κύριε Σβάμπ δεν πρόκειται να σας περιορίσω διότι έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την ε, ενδιαφέρουσα εισαγωγή. Νομίζω ότι επειδή την προηγούμενη φορά ήμουν σύντομο, τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στα θέματα τα οποία δεν έθιξα την προηγούμενη φορά. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σημερινή συνεδρίαση, η οποία εκπροσωπείται με ε, μία ευρεία πληθώρα συνεργατών, κατά τρόπον ώστε να μπορέσει να μας διευκολύνει σαν Ευρωβουλευτές και να καταλάβουμε μέσω των απαντήσεών τους για τις συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες έχουν διατυπώσει στην οδηγία. Ευχαριστώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σχετικά με το Συμβούλιο, το οποίο δεν ήρθε στην τελευταία συζήτηση καθόλου, ο κύριος Ντόλινγκ είναι διαθέσιμος ανα πάσα στιγμή ε, για ερωτήσεις, οπότε θέλω να ευχαριστήσω την Σουηδική Προεδρία, η οποία κάνει ε, πολύ σοβαρές προσπάθειες για να προχωρήσει αυτός ο φάκελος και ε, θα ήθελα ε, εφόσον έχω ευχαριστήσει ήδη την προηγούμενη φορά την σκιώδη συγγήτρια να μην το πράξω και τώρα. Αντιθέτως όμως θα ήθελα να σας πω τι γνωρίζω, ποιες είναι οι πληροφορίες που έχω, διότι μετά από πάρα πολλές συζητήσεις ε, με οργανώσεις για την προστασία των καταναλωτών, για διάφορου, με διάφορους εκπροσώπους. Σήμερα ήρθε η, ε, η υπουργό της Φιλανδίας, η οποία μας πρότεινε διάφορες λύσεις, η οποία όμως ε, συγχρόνως συνεπάγεται και ορισμένα προβλήματα νέα και δεν βλέπω πού θα καταλήξουμε. Όπως όμως είπε και σήμερα το πρωί η κυρία Γκέπχαρτ, είμαι αντίθετο στην πλήρη εναρμόνιση και αυτό θέλω να το τονίσω καταρχήν. Διότι ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συμφώνησε με την ε, πρόταση της Επιτροπής για την συνθήκη της Ρώμης 1 ε, η οποία πρέπει να ισχύσει από τις αρχές του 2010 και θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα που δεν έχουμε εξετάσει επαρκώς μέχρι στιγμής και γι' αυτό η συζήτησή μας πρέπει να ολοκληρωθεί πριν ισχύσει αυτή η αλλαγή. Μετά πρέπει ε, να δούμε ε, τι έχει γίνει με την απόφαση Alpenhood που είναι ένα αυστριακό ξενοδοχείο το οποίο προσφέρει ε, υπηρεσίες στους πελάτες του και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεώρησε ότι αφού η προσφορά αυτή ε, οφείλεται, ε, έχει διαδοθεί στο διαδίκτυο μπορεί να προσελκύσει και ε, αλλοδαπούς πλέον των αυστριακών δυνητικών πελατών πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να ισχύσουν οι, οι ρήτρες προστασίας των καταναλωτών των κρατών αυτών και όχι μόνο η αυστριακή πράγμα που θα, έλεγε, θα εννοούσε το ξενοδοχείο Alpenhut πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις προστασίας ε, καταναλωτών για 27 χώρες αντί για μόνο μία. Ε, και ε, από 1η Ιανουαρίου η αναδιατυπωμένη οδηγία θα επηρεάζει και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αναφερόμαστε λοιπόν καταρχήν στα δικαιώματα των καταναλωτών πριν την απόφαση για το ξενοδοχείο Alpenhut και ε, η σημερινή ελάχιστη εναρμόνιση ε, αναφέρεται στο κεφάλαιο 4 και ε, έχει λειτουργήσει. Αλλά όσον αφορά ε, ε, τις περαιτέρω διατυπώσεις ε, θα μπορεί κάθε κράτος να αναλάβει και ευρύτερες καλύψεις στα πλαίσια αυτής της οδηγίας. Έχουμε δηλαδή προς το παρόν ένα σύστημα έξι μηνών για αντίδραση και δύο ετών εγγύσεως και εγώ είδα ότι νομικά ότι αυτή η σωστή εφαρμογή ε, τελικά δεν ισχύει ε, στην πράξη ε, στον εμπορικό κόσμο διότι αγόρασα ε, μια εξαιριστική μηχανή μετά από ε, τρεις εβδομάδες ειδοποίησα τον πολιτή ότι δεν λειτουργούσε και μου είπε δεν μπορώ να κάνω τίποτα πρέπει να απευθυνθείτε στο κατασκευαστή. Λοιπόν, δεν είχα ασχοληθεί ε, με αυτή την οδηγία οπότε μετά ήρθα σε επαφή με ε, το εργοστάσιο και μετά ε, επανήλθα στον ε, πολιτή, στο έμπορο, ο οποίος μου είπε ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι αυτό θα έπρεπε να παίρνει πίσω τα, τις μηχανές οι οποίες χάλασαν μέσα στην περίοδο της εγγύσεως. Δηλαδή, όπως είπε η κυρία Κούνεβα, υπάρχουν θέματα τα οποία καταναλωτές πρέπει να ε, λύσουν πολύ καλά και πρέπει να δούμε αν πρέπει απλώς να εστιαστούμε στο ουσιαστικό κείμενο ή πρέπει να επιλύσουμε τα θέματα που προκύπτουν από τα δικαιώματα των καταναλωτών. Διότι η εναρμόνιση έχει νόημα μόνο αν υπάρχει πλήρης εναρμόνιση. Αλλά η εναρμόνιση αυτή ουσιαστικά αναφέρεται σε έναν μικρό τομέα της νομοθετικής εξελίξεως η οποία διαδραματίζεται κατά την διεξαγωγή μιας και αγοράς διότι ε, δεν ε, παρακολουθείτε το τι πρόκειται να συμβεί κατόπιν, ε, τι μπορεί να έχει συμβεί μέχρι τη στιγμή της πωλήσεω και έτσι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία μιλά για πλήρη εναρμόνιση δεν επιλύει όλα τα νομοθετικά προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν στα πλαίσια της εγγύησεως. Πιστεύω λοιπόν ότι ένα από τα, τους στόχους τους οποίους επιζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την εναρμόνιση φτάνει στην υπερβολή. Και γι' αυτό θα ήθελα τώρα να ε, σκιαγραφίσω διάφορα θέματα που με απασχολούν ιδιαίτερο στο τέταρτο κεφάλαιο. Καταρχήν, προτού αναφερθούμε στην πλήρη εναρμόνιση και η κυρία Γκέπχαρτ πολύ σωστά είπε την προηγούμενη φορά διότι δεν μπορούμε να, ε, ότι δεν μπορούμε να το εξετάσουμε εξαντλητικά. Ε, το πρώτο θέμα είναι ποια είναι η σωστή λύση η οποία καταρχήν θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών και από την άλλη πλευρά ε, θα μπορεί να εξασφαλίσει στον έμπορο ή στον κατασκευαστή ε, την δυνατότητα να έχει ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς μέσα στην ενιαία αγορά. Και εδώ θα αναφερθώ σε ορισμένα συγκεκριμένα θέματα. Πρώτον, εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στην παράδοση του προϊόντος, του εμπορεύματος, διότι λέγεται ότι θα πρέπει να έχει παραδοθεί το εμπόρευμα εντός 30 ημερών. Ο, ε, ο έμπορος ε, θα πρέπει να έχει παραδώσει το εμπόρευμα εντός 30 ημερών ε, για κάποιο εύλογο λόγο. Διαφορετικά θα εξαντλούσε κάθε φορά ο έμπορος 30 ε, δεν πρέπει δηλαδή να φταίει ο έμπορος για τις καθυστερήσεις ε, αλλά εδώ μας παραπέμπουν εις ε, την οδηγία για την παροχή υπηρεσιών η οποία αναφέρεται σε διαφορετικές διατάξεις. Μετά, ε, στο κεφάλαιο 4 μπορούμε να περιλάβουμε διάφορες, νομοθετι... Ε, διάφορες νομοθετικές διατάξεις, αλλά δεν πρέπει εδώ οι διατάξεις αυτές να είναι σε αντίφαση με αυτή των ταχυδρομικών υπηρεσιών, παραδείγματο χάρη. Στο άρθρο 23 είναι ασαφές ποιος είναι υπεύθυνος αν ο πολιτής έχει παραδώσει σε ένα μεταφορέα το εμπόρευμα και το εμπόρευμα μπορεί να πάθει μια ζημιά κατά τη μεταφορά. Αυτές είναι ασάφειες οι οποίες θα πρέπει επίσης να διευκρινιστούν. Μετά, το θέμα ε, της ε, δυνατότητας ε, άμεσης επιστροφής, δηλαδή right to reject, όπως λέγεται αγγλικά. Σύμφωνα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το σχέδιο της οδηγίας βασίζεται στην αρχή της πλήρης εναρμονήσεως αλλά οι γενικές ε, συμβατικές διατάξεις ε, ε, αποκλείονται εφόσον αναφέρονται στο εμπορικό δίκαιο και άρα η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το right to reject δεν είναι αυτή που υπάρχει στην Αγγλία αλλά διαφορετική και ξέρω ότι αυτό συνεπάγεται διάφορα προβλήματα διότι οι χώρες οι οποίες έχουν ε, την διάταξη right to reject δεν θέλουν να την ε, εγκαταλείψουν και ε, δεν θέλουμε ούτε εμείς στην Ευρώπη να μειώσουμε τα δικαιώματά μας πρέπει όμως να συζητήσουμε αν το right to reject δηλαδή το δικαίωμα απορρίψεως είναι ένα προσόν για τον καταναλωτή στην Ευρώπη διότι θα θέλαμε τα νέα δικαιώματα που θα υπάρχουν να μπορέσουν να ενταχθούν ενταχθούν επικοδομητικά στην ένωμη τάξη και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση τίνει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων είναι πολύ ουσιαστικό θέμα. Θα πρέπει όμως το εμπόριο να μπορεί να λειτουργήσει ε, σωστά ε, μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών αρχών ε, και να εφαρμόσουμε την αρχή Pacta Sunt Servanda. Και αυτή η αρχή θα πρέπει να παραμείνει σεβαστή. Στην αρχή η Σουηδική η Σουηδική Προεδρία είχε προτείνει ότι το right to reject θα πρέπει να ισχύσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις πρώτες 14 μέρες αλλά μετά καταλήξαμε σε μια συμβιβαστική πρόταση η οποία ε, θέλει να αποφύγει τις καταχρήσεις του δικαιώματος και γι' αυτό το κεφάλαιο 4 θα πρέπει να διατυπωθεί με πολύ προσεκτικό τρόπο διότι αν ε, πρόκειται, μία εστιασμένη, πρόκειται για μια ε, εστιασμένη εναρμόνιση κάποιου τομέα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το διευκρινίσει για να αποφύγουμε ε, να ε, να επηρεαστούν οι εμπορικές ε, συνήθειες οι οποίες υπάρχουν και κατοχυρώνται νομικά σε διάφορα κράτη. Μετά, το βάρος της απόδειξης, το οποίο ε, επεκτείνεται για 10 χρόνια. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος αγόρασε ένα εμπόρευμα, 10 χρόνια μετά την αγορά θα έχει το δικαίωμα να αποδείξει ότι το εμπόρευμα τη στιγμή που του παραδόθηκε είχε ένα, μια ζημιά η οποία αποκαλύφθηκε μετά από 10 χρόνια. Πιστεύω ότι αυτό θα επιτευχθεί μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, θα συνεπάγεται φοβερές δαπάνες για τον καταναλωτή. Υπάρχουν όμως προϊόντα τα οποία ε, επιβάλλουν να υπάρχει μία τέτοια λύση αλλά αυτά θα πρέπει να επιλύονται σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή τα δέκα χρόνια αυτά δεν θα μπορούν να ισχύσουν για, τις, ε, για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και ε, χρειάζεται ακόμη να μελετηθεί το θέμα. Και τέλος όσον αφορά το, ε, την αρχή της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πει, θεωρεί ότι ο κατασκευαστής πρέπει να επιλέξει τον τρόπο επιδιορθώσεως και όχι ο καταναλωτής. Εγώ όμως πιστεύω ότι εδώ θέλει σκέψη, διότι το πλαίσιο αναφοράς δημιουργεί ένα δικαίωμα εγγύησης και αυτά θα πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τέλος, ολοκληρώνοντας αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι ακόμη και σε τμήματα του κεφαλαίου 4 υπάρχουν δυνατότητες βελτιώσεως αλλά θα πρέπει να επιζητήσουμε σωστές λύσεις ώστε να προστατεύουμε αφενός των καταναλωτών αλλά να μπορούμε να διεκπεραιώνουμε και ενιαία το διασυνοριακό το διασυνοριακό εμπόριο στα πλαίσια της αποφάσεως για το ξενοδοχείο Alpenhood. Θα ήθελα πέραν όμως της παρουσιάσεώς μου να ευχαριστήσω την γραμματεία της Επιτροπής και ιδίως τον νέο γραμματέα ο οποίος από 1η Δεκεμβρίου αντικατέστησε τον προηγούμενο και προσβλέπω στη συζήτηση που θα κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σουάμπ για την εξαιρετική σας παρουσίαση και για τα ιδιαίτερως ενδιαφέροντα θέματα τα οποία παρουσιάσατε και τα οποία ασφαλώς θα συζητήσουμε τώρα με μεγάλο ενδιαφέρον. Θα δώσω τώρα το λόγο στον σκιώδη συγητή, την κυρία, στη σκιώδη συγητή, την κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητή Μπερναντέτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σουάμπ για αυτή την ε, εισαγωγή και επίσης για την καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα και που υποθέτω ότι θα συνεχιστεί και μελλοντικά. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με μια από τις πρώτες παρατηρήσεις που κάνατε, την εφαρμογή του δικαίου στην Γερμανία. Αυτό είναι ένα θέμα, το ότι πρέπει να γίνεται η εφαρμογή ένα προς ένα, όπως ε, λένε πάντοτε οι χριστιανοδημοκράτες, ενώ εμείς οι χριστιανοδημοκράτες θεωρούμε ότι μπορούμε να το ξεπεράσουμε ή να προσαρμοστούμε στην εκάστοτε παράδοση. Γιατί το ευρωπαϊκό δίκαιο δίνει τέτοιο περιθώριο προσαρμογής εκεί που κρίνεται αυτό λογικό. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια, ένα πρώτο, μια πρώτη ενδοκερμανική διένεξη. Τώρα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την σύνοψη, η οποία είναι ιδιαίτερως ε, χρήσιμη. Εγώ κοίταξα εδώ και εκεί τις οδηγίες. Ε, είναι πολύ χρήσιμο όταν ε, μπορεί να τις εξετάσει κανείς όλες σε μια τέτοιου είδους σύνοψη. Θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμη επίσης η δεξιά στήλη εκεί όπου αναγράφονται τα σχόλια. No chance γράφει το κείμενο. Ε, αλλά μόνο εφόσον παραλείψει κανείς ε, το άρθρο 4. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια σημαντική διάκριση. Στο αρχικό κείμενο το θέμα ήταν η ελάχιστη εναρμόνιση την οποία μπορούσαν να ξεπεράσουν οι χώρες μέλη εφόσον το επιθυμούσαν, ενώ τώρα στο παρόν κείμενο προβλέπεται μια πλήρης εναρμόνιση, δηλαδή δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτή την ανάγκη εναρμόνιση οι χώρες μέλη και αυτό είναι μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο κειμένων και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να το παραβλέπει κανείς όταν εξετάζει αυτή τη σύνοψη. Δεν θα πρέπει δηλαδή να το αφήσουμε κατά μέρος. Ε, και εδώ έρχομαι στην ε, βασική μου εκτίμηση κύριε Σβάμπ, όπου σας είπα δεν συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι μπορούμε να συζητήσουμε κεφάλαιο προς κεφάλαιο και να αφήσουμε το άρθρο τέσσερα κατά μέρο. Κύριε Σφαμπ, δεν συμφωνώ μαζί σα. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται, γιατί οι συνέπειε πραγματικά είναι εξαιρετικά σημαντικέ. Εάν στο ευρωπαϊκό δίκαιο προβλέπεται πράγματι μια πλήρη εναρμόνιση στον τομέα αυτό, κατά το οποίο δεν ελπίζω και πραγματικά θα το πολεμήσω, τότε θα πρέπει να υπάρξουν εντελώς διαφορετικές τροπολογίες από αυτές που αναφέρονται στην ελάχιστη εναρμόνιση. Αν θέλετε οπωσδήποτε να έχετε την πλήρη εναρμόνιση και είπατε ο ίδιος ότι σε αυτό το κεφάλαιο πραγματικά εσείς ο ίδιος αντιφάσκετε. Ε, ε, ε, τότε θα πρέπει να το μπορούν να το αποφασίσουν οι ίδιες οι χώρες. Μόνο τότε μπορώ να το σκεφτώ. Αλλά δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήταν πρόθυμη να κάνει κάτι τέτοιο. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε ποιες ακριβώς είναι οι συνέπειες. Ε, και τώρα έρχομαι στο κεφάλαιο 4, ε, τομέας εφαρμογής, άρθρο 21. Εδώ περιορίζεται στα είδη, στα εμπορεύματα. Και νομίζω ότι θα ήταν καλό να κάνουμε και κάποια σκέψη σχετικά με τις υπηρεσίε, όχι μόνο με τα είδη. Γιατί εδώ και 30 ή 40 χρόνια ήταν πάντοτε το θέμα των υπηρεσιών αυτό το οποίο παραλείπαμε. Αλλά βεβαίως κάποτε τα προβλήματα γίνονται τόσο οξέα που νομίζουμε ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με μια τέτοια μεγάλη επίθεση, πράγμα που όμως στην ουσία μας φέρνει προς τα πίσω όσον αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τώρα, ε, το άρθρο 3 δεν ισχύει για τα ανταλλακτικά. Ε, νομίζω ότι είναι εντάξει, θα μπορεί, μπορεί να το διατυπώσει κανείς. Αλλά τι, γίνεται με την ε, προθεσμία που προβλέπετε. Αν για παράδειγμα στο πλυντήριό μου ε, τα φτύσει το ε, μηχάνημα, η μηχανή, ε, ένα πλυντήριο που αγόρασε πριν από έξι μήνες. μπορούμε να βάλουμε ένα καινούριο κινητήρα, μια καινούρια μηχανή. το πλυντήριο λειτουργεί ε, μερικούς μήνες ακόμα και στη συνέχεια ξαναχαλάει. Συνήθως ε, υποθέτει κανείς ότι ε, η ζωή ενός τέτοιου κινητήρα είναι κάπως μακρύτερη. Αλλά δεν προβλέπεται όμως κάτι τέτοιο, μια τέτοια προθεσμία, γιατί το μηχάνημα συνολικά, το πλυντήριο συνολικά είναι πολύ παλαιότερο, είναι πλέον 3,5-3 ετών. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω τι γίνεται με τα ανταλλακτικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ε, προθεσμία, μια εγγύηση λειτουργίας των ανταλλακτικών. Τώρα, έχουμε το άρθρο 22. Νομίζω ότι το σημείο 2 είναι σωστό συμφωνώ να πούμε ότι η απέτηση του καταναλωτού για αποπληρωμή όλων των υπηρεσιών μέσα σε 7 μέρες από την στιγμή της παράδοσης. Αλλά τι σημαίνει ε, στιγμή, ε, ημερομηνία παράδοσης. Νομίζω ότι ε, αυτό κάνει τα πράγματα πολύ πολύπλοκα. Δηλαδή η ιδιοκτησία του καταναλωτού ε, Δηλαδή τι γίνεται αν για παράδειγμα εγώ έχω πάει διακοπές μια εβδομάδα και η παράδοση γίνεται σε ένα γείτονα σε ένα φίλο και χαλάει το μηχάνημα. Ε, τι γίνεται όταν ισχύει αυτή η προθεσμία των 7 ημερών στην περίπτωση αυτή. Νομίζω ότι θα πρέπει να το διατυπώσουμε κάπως πιο προσεκτικά, γιατί αυτό είναι εις βάρος τελικά του εμπόρου, αυτού που παρέδωσε το, τη συσκευή. Βλέπετε, δεν σκέφτομαι μόνο το όφελος του καταναλωτού, αλλά στην περίπτωση αυτή και του επιχειρηματία. Τώρα, όσον αφορά την ε, μεταφορά των κινδύνων, νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχει κάποιος κίνδυνος απώλειας ή ζημίας ε, κατά την παράδοση. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Ε, νομίζω είναι αυτονόητο και ήταν σωστό πάντα μέχρι τώρα. Αλλά στο πλαίσιο αυτό δεν καταλαβαίνω πολύ καλά το σημείο 2. Ίσως θα μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας διευκρινίσει το σημείο αυτό. Πώς πρέπει να το καταλάβουμε δηλαδή, να το διαβάσουμε. Τι γίνεται. Και παίρνω πάντα, πάλι το παράδειγμα ότι εγώ είμαι σε διακοπές και παραδίδεται η συσκευή στο γείτονα που δεν τον έχω επιφορτήσει, αλλά το ταχυδρομείο του το παραδίδει γιατί αυτός έτυχε να βρίσκεται εκεί. Τι γίνεται λοιπόν στην περίπτωση αυτή όταν εγώ δεν μπορώ να κάνω τα αναγκαία διαβήματα που προβλέπετε για να αποκτήσω καταρχήν την κυριότητα του είδος και μετά να υποβάλω τις αξιώσεις μου. Τι συμβαίνει λοιπόν για αυτό το διάστημα. Ε, είναι ο γείτονας υπεύθυνο σε αυτό το μεσοδιάστημα που εγώ λείπω. Ε, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα πρέπει να μας το διευκρινίσετε. Δεν είμαι νομικός ε, και ίσως η αλήθεια κρύβεται σε κάποιες ε, λεπτομέρειες που εγώ δεν τις γνωρίζω, αλλά θα πρέπει νομίζω να διαλευκανθούν. Γιατί δεν είναι δυνατόν να παρακαλέσω το γείτονά μου να αποδεχθεί επισήμως κάτι εκ μέρους μου. Ε, εγώ είμαι υπεύθυνη να το κάνω. Τώρα, όσον αφορά την ε, συμφωνία με την σύμβαση. Στο σημείο 2 αναφέρονται διάφοροι λόγοι ε, κατά πόσο πληρούνται όλες οι διατάξεις της σύμβασης, του συμβολέου μάλλον, η συμφωνία με το συμβόλαιο, η συμβατότητα με το συμβόλαιο. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες χώρες μέλη που θέτουν κάποιους επιπλέον όρους και που θα πρέπει να καταργηθούν εάν ισχύσει το άρθρο 4, δηλαδή η πλήρη εναρμόνιση. Και με τον τρόπο αυτό επέρχεται μια επιδείνωση στα δικαιώματα των καταναλωτών σε αυτές τις χώρες μέλη όσον αφορά αυτές τις ε, διατάξεις. Στο άρθρο 24, σημείο 3. Εάν δεν υπάρχει παραβίαση του συμβολέου, ε, εφόσον υπάρχει, ε, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής γνώση ε, για την ε, παραβίαση, για τυχόν παραβίαση του συμβολέου. Δεν ξέρω, διατυπώνεται το, ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει σαφή γνώση για τυχόν παραβιάση του συμβολέου. Τι σημαίνει αυτό, είναι τελείως αόριστη αυτή η διατύπωση και εδώ παίζει και ένα ρόλο το λεγόμενο φορτίο της απόδειξης, το βάρος της απόδειξης Δηλαδή, ο καταναλωτής θα έπρεπε να είναι σε γνώση για τυχόν παραβιάση κλπ, αλλά ίσως δεν ενημερώθηκε, δεν διάβασε τα email του, δεν ξέρω. Ε, τι, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Αυτά είναι θέματα τα οποία ανακύπτουν και τα οποία θα ήθελα να διευκρινίσω. Και στο σημείο 4, εδώ διαρωτώ με, τι εννοεί το σημείο γάμα ο επαγγελματίας ο οποίος δεν είναι δεσμευμένος στις ε, επίσημες ε, δηλώσεις του, στις δημόσιες δηλώσεις τους, εάν η απόφαση αγοράς ε, δεν επηρεάζεται από αυτές τις δημόσιες δηλώσεις του εμπόρου. Τι σημαίνει αυτό. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εάν έχει ο έμπορος κάποιες ε, πληροφορίες, αυτό είναι καθοριστικό για την αγορά του προϊόντος, όχι. Τι εννοείται με αυτό. Είναι καθοριστικό ή δεν είναι καθοριστικό για την ε, απόφαση αγοράς του προϊόντος. Δεν καταλαβαίνω. Νομίζω θα πρέπει να διευκρινιστεί. Γιατί ε, δεν ξέρω πώς θα πρέπει να το ερμηνεύσουμε. Ε, και βλέπω να ανέβει ο κύριος Σβάμπ. Προφανώς ε, έθεσε και ο ίδιος τον εαυτό του αυτά τα ερωτήματα. Και συνέχεια έχουμε το άρθρο 25, το οποίο για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό. Ο έμπορος έχει την ευθύνη για κάθε παραβίαση του συμβολέου ε, κατά το διάστημα της ε, παράδοσης του προϊόντος στον καταναλωτή. Τι σημαίνει παραβιάσεις του συμβολέου. Πρόκειται για την ευθύνη, για την τήρηση των προθεσμιών, αλλά και από πότε ισχύει η αντιστροφή, η λεγόμενη αντιστροφή του βάρους της απόδειξης στο άρθρο 28, δηλαδή μέσα σε έξι μήνες εφόσον μεταφερθεί μετά τη μεταφορά του κινδύνου ε, στον ε, αγοραστή, ζητώ συγγνώμη από τις διερμηνείς λέει η ομιλήτρια, ε, εάν υπάρχει υπόνοια ότι υπάρχει παραβίαση του συμβολέου την εποχή της ε, μεταφοράς του κινδύνου και για ένα διάστημα έξι μηνών. Δηλαδή για τους έξι μήνες δεν ισχύει η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, αλλά μετά την ε, παρέλευση των έξι μηνών ισχύει η αρχή της αντιστροφής του βάρους της απόδειξης. Και διερωτώμε κατά πόσο αυτό είναι αποδεκτό. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ζητήσει σχετικά ε, συχνά σε σχέση με το θέμα της ασφαλείας των προϊόντων, όπου είπατε ότι δεν ήταν να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο σκηνοβούλιο. γιατί ακριβώς εκεί όπου πρόκειται για κάποια προϊόντα τα οποία είναι πιο πολύπλοκα, ο καταναλωτής δεν έχει απολύτως καμία δυνατότητα να αποδείξει πού και γιατί υπάρχει κάποιο λάτωμα στο προϊόν ε, γιατί υπάρχει αυτό το ελάττωμα, η ζημία, ενώ βεβαίως οι κατασκευαστές έχουν κάθε δυνατότητα να ελέγξουν πού εντοπίζονται τα ελαττώματα των προϊόντων τους. Συνεπώς λοιπόν ε, νομίζω ότι αυτή η αντιστροφή του βάρους απόδειξης ε, δεν θα πρέπει να ισχύει. Νομίζω θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να την αμφισβητήσουμε αυτή την αρχή. Τώρα, ανακύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα και Τώρα θα περάσω στις εγγύσεις εκ μέρους των κατασκευαστών. Ε, και εδώ με έχουν καταπλήξει δύο σημεία. Αναφέρεται ότι η δήλωση ε, ότι η εγγύηση περιλαμβάνει τα εξής. Δηλαδή, η εγγύηση δεν μπορεί να μεταφερθεί σε έναν μεταγενέστερο αγοραστή. Τρία, παράγραφος 3.1. Λοιπόν, εδώ λέει το δικαίωμα του καταναλωτή να μεταπολίσει το είδος ε, συνοδεύεται από ένα περιορισμό τις ε, εγγύηση. Στη μία διάταξη δεν μπορεί η εγγύηση να μεταφέρεται στον επόμενο ε, αγοραστή. Ε, από την άλλη υπάρχει μια διαταξη δεν μπορει η εγγυηση να μεταφερεται στον επομενο αγοραστη απο την αλλη υπαρχει μια ρήτρα που αναφέρεται στην μη κακή χρήση του ε, συμβολέου. Σημείο 3 του άρθρου 29. Κατόπιν επιθυμίας του καταναλωτού, ο κατασκευαστής ε, ε οφείλει να θέσει στη διάθεσή του την εγγύηση ε, τι θα πρέπει να γίνει όταν ο κατασκευαστής δεν μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει εγγύηση για ένα προϊόν. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκέπχαρτ για αυτές τις ε, διευκρινήσεις και αυτά τα ερωτήματα. Ε, το θέμα είναι ιδιαίτερο τεχνικό. Μήπως ο σκιώδης εισηγητής ο κύριος ε, Μάντες, ο η κυρία Τουρενέν, ο κύριος Μπίλεν και ο κύριος Τρενταφυλλίδης έχουν κάποια αντίρρηση στο να πάρει το λόγο ο κύριος Σαμπάτ γιατί χτύπησε το πόδι του δυστυχώς και πρέπει να φύγει κατεπηγόντως για τη Γαλλία. Νομίζω ότι δεν έχει κανείς καμία αντίρρηση. Κύριε Αμπάντ, ε, έχετε το λόγο και σας ευχαριστούμε που παρά το δραματισμό σας ε, ήρθατε εδώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και σε εσά τους ε, συγητές και σχεδόν συγητές που με επιτρέπετε να παρέμβω. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ανδρέα Σβάμπη για την ποιότητα της εργασίας του. Έχει μεγάλες ικανότητες ε, ε, διαβούλευσης και συνεργασίας. Ε, έτσι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την προστασία του καταναλωτή, εγγυόμενη την ε, νομική σταθερότητα των εταιριών μας, καθώς και την οικονομική τους άνθηση. Σήμερα μιλάμε για το κεφάλαιο 4 που έχει σχέση με τα δικαιώματα του καταναλωτή και με τις ε, συμβάσεις πωλήσεων νομικές εγγυήσεις και ιδιαίτερα ευθύνη για την ε, περίπτωση ε, βλάβης η έλλειψη συμμόρφωση. Ε, προβλέπεται μια εγγύηση για δύο χρόνια, δηλαδή από τη στιγμή που ο καταναλωτής ε, παίρνει αυτά τα αγαθά, έχει δύο χρόνια εγγύηση Στη Γαλλία με ειδοποίησαν διάφορες ε, νόσες Γάλλων καταναλωτών και είναι αλήθεια ότι κάποια ερωτηματικά προκύπτουν εδώ. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι τι θα γίνει αν ένας καταναλωτής αγοράσει για παράδειγμα ε, πλακάκια κατά του, που, που είναι ανθεκτικά υποτίθεται στον πάγο και τα δύο πρώτα χρόνια περάσει τους χειμώνες ε, χωρίς πρόβλημα και το τρίτο χρόνο ε, παρουσιαστεί πρόβλημα. Ε, μια τέτοια περίπτωση δεν εμπίπτει στο σχήμα που μας παρουσιάζει η Κομισιόν. Είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα για τους Γάλλους καταναλωτές που αυτή τη στιγμή χαίρουν ενός συστήματος πιο προστατευτικού από αυτό που προβλέπεται στο πλαίσιο αυτής της πρότασης. Βεβαίω, στόχο μα δεν είναι να διατηρήσουμε όλα τα εθνικά δικαιώματα σε θέματα προστασία του καταναλωτή, αλλά αντίθετα, όπω είπαμε, να προχωρήσουμε προ μια στοχευμένη εναρμόνιση. Αλλά χρειάζεται να έχουμε τέτοια συγκεκριμένα παραδείγματα που δείχνουν ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη μπορεί να προκύψει ένα αίσθημα φόβου ε, σε σχέση με ένα κεκτημένο δικαίωμα. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για αυτά τα θέματα και για την αντιπροσωπεία του ΕΛΚ, του, τη, τη γαλλική αντιπροσωπεία του ΕΛΚ, μπορώ να σα πω ότι συνάντησα και άλλου συναδέλφου που μοιράζονται τις ίδιε ανησυχίες και μάλιστα ε, το κοινοβούλιο μα πριν από λίγε μέρε ανακοίνωσε μια έκθεση για αυτό το θέμα και οι επιφυλάξει είναι πολύ έντονε όπω διαπιστώνουμε μετά από ανάγνωση της έκθεσης αυτής. Εργασία που γίνεται λοιπόν σήμερα εδώ, το θέμα του πιθανού κινδύνου ή του ενός κρυφού ελαττώματος και καλυμμένου ελαττώματος είναι ουσιώδης εδώ. Θα πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί αυτή η οδηγία ανάλογα με το συγκεκριμένο σημείο γιατί είναι προς το συμφέρον μας ως Ευρωπαίοι εκπρόσωποι ε, να μπορέσουμε να επιτρέψουμε σε όλους να κατανοήσουν ε, τα διακυβεύματα αυτής της οδηγίας και να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε όπως αυτό που σας ανέφερα μόλις τώρα. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει η κυρία Τούρινεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μου χρειαστεί ίσως κάποιος χρόνος, ίσως να μην μακρηγορήσω όσο οι άλλοι, αλλά έχω κάποιες παρατηρήσεις ωστόσο να διατυπώσω. Και κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε σήμερα εδώ αυτά τα θέματα, όπου στο, και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 4, όπου προσπαθούμε να συγκρίνουμε αυτό το πίνακα, όπου βλέπουμε τις διαφορές ανάμεσα στο τι είχαμε πριν. Είναι αλήθεια πως υπάρχουν πολλές αλλαγές ε, και μη σημαντικές αλλαγές, αλλά εγώ πιστεύω πως είναι πραγματικά

σημαντικό γιατί υπάρχουν αλλαγέ οι οποίε θεωρούνται μη σημαντικέ, ενώ είναι. Θα σα δώσω παραδείγματα γιατί έχουμε όλοι σε διάφορε χώρε πιο ευνοϊκού κανόνε από αυτού που βλέπουμε εδώ στην οδηγία και σύμφωνα με αυτήν δεν θα μπορούσαμε να τα διατηρήσουμε. Για το πεδίο εφαρμογή εγώ δεν καταλαβαίνω ακριβώ ε, τι συμβαίνει γιατί στο κεφάλαιο 1 λέγεται πω η οδηγία αυτή θα ισχύσει για τα εμπορεύματα και για τι υπηρεσίε. ενώ στο κεφάλαιο 4 δεν είναι πλέον τόσο Μας λέει ότι όταν πρόκειται για έναν μεικτό στόχο, γιατί θα μπορούσαμε ας να έχουμε ένα εμπόρευμα και μια ε, υπηρεσία ταυτόχρονα, τότε η οδηγία δεν ισχύει παρά μόνο για το εμπόρευμα. Μα τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Για παράδειγμα, αν πρέπει να τοποθετήσω πλακάκια σπίτι μου η οδηγία αυτά με καλύπτει μόνο για τα πλακάκια και όχι για τον τρόπο με τον οποίο ε, τοποθετούνται. Και αν για παράδειγμα πάω στο κομμωτήριο για να βάψω τα μαλλιά μου και αρχίσουν να πέφτουν τα μαλλιά μου, εκεί τι ακριβώς θα ισχύσει. Θα πρέπει λοιπόν ακριβώς να ορίσουμε τι εννοούμε εμπόρευμα και τι εννοούμε υπηρεσία. Βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία συνδέονται. Ε, σε σχέση με τους ε, συμβατικούς κανόνες. Έχουμε ήδη ε, εξετάσει το θέμα και στο παρελθόν και γίνεται πολύ περίπλοκο το θέμα γιατί ορισμένες φορές έχουμε διάφορα στοιχεία που αναμειγνύονται και θα ήθελα να προσπαθήσω να θίξω ορισμένα, να αναφέρω μάλλον συγκεκριμένα άρθρα. Η κυρία Γκέπαρντ ήδη μίλησε για το 21.3, για τα ανταλλακτικά και έχουμε και ένα άρθρο σε σχέση με την παράδοση αγαθών και λέει ότι 30 μέρες ε, το αργότερο μετά από τη σύναψη της συμφωνίας θα πρέπει να γίνεται η παράδοση. Αλλά εδώ αν δούμε μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία υπάρχουν ε, συμβόλαια που πρέπει να εκτελεστούν άμεσα και θα μπορούσαμε να διερωτηθούμε τι γίνεται εδώ με τα ποσά που κατατίθενται κατά τη διάρκεια της σύναψης της συμφωνίας. Υπάρχουν όμως πολλές χώρες, όπως η Ισλανδία, η Δανία και η Σουηδία, που έχουμε διαφορετικούς κανόνες εφόσον πρόκειται για εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για ίδια κατανάλωση. Έχουμε προβλήματα επίσης στις τι συσκευασίε. Ε, παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου. Ο καταναλωτής πρέπει να δει αν θέλει μείωση της τιμής, έκπτωση ή αν θέλει αλλαγή ενός ελαττωματικού προϊόντος, αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα ο πολιτής αποφασίζει. Εγώ πιστεύω πως ο καταναλωτής είναι αυτός που πρέπει να προστατευτεί και αυτός που μπορεί να επιλέξει. Αυτό που έχουμε εδώ είναι απαράδεκτο. Και Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι που συμφωνούν μαζί μου. Άρθρο 26, παράγραφος 3 ε, μέχρι 5 εδώ έχουμε τη δυνατότητα για την επισκευή ενός προϊόντος. Έχουμε κάποιες φορές εδώ και αντικατάσταση του προϊόντος που προτείνεται, αλλά εμείς είμαστε κατά ως πράσινοι, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα πλήρη εναρμόνιση. Πιστεύουμε πως ο καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να καταργήσει τη συμφωνία αν το εμπόρευμα ήταν ελαττωματικό εξ αρχής θα πρέπει να είναι δυνατόν σε εθνικό επίπεδο να υπάρχει σεβασμός ε, των ε, δικαιωμάτων του καταναλωτή και συζήτησε το θέμα με την Επιτροπή και από ό,τι κατάλαβα δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα να μπορεί κανείς να διατηρήσει το δικαίωμα απόρριψης του το right to reject στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν καταλαβαίνω όμως πώς κάτι τέτοιο θα είναι δυνατόν. Δηλαδή, συμβατικές ε, διατάξεις σε εθνικό επίπεδο ε, έρχονται σε αντίθεση με αυτή την οδηγία. Γιατί εδώ μας προτείνεται κάτι διαφορετικό. Γιατί να έχουμε εδώ κάτι διαφορετικό στα κράτη-μέλη. Και στο άρθρο 26 παράγραφος 3 υπάρχουν ένα σωρό διατάξεις. Τι θα είναι δυνατόν, τι θα μπορούμε να κάνουμε και πώς θα προχωρήσουμε. Εδώ κάτι μου διαφεύγει. Δεν βλέπω πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε το right to reject με βάση το ε, τωρινό κείμενο. Άρθρο 28 παράγραφος ε, 1 η διάρκεια δύο ετών για ε, καταγγελία ή για επιστροφή. Αυτή είναι η ελάχιστη χρονική περίοδος, αλλά αυτό μπορεί να παρουσιάζει επιδείνωση της κατάστασης για τη Γερμανία ή το Βέλγιο, γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες όπου το δικαίωμα αυτό μπορεί να ξεπερνά τα δύο χρόνια. Και Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τον πίνακα αυτό, γιατί εδώ δεν αναφέρω, λέει ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές, αν και είναι αντίθετο, περνάμε από το μήνυμο στο μάξιμο. Η Δανία, η Ισλανδία, Γαλλία, κάτω χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, στι χώρες αυτές σήμερα μπορεί κανείς να έχει μεγαλύτερη χρονική περίοδο από αυτή που προτείνεται γιατί εδώ δεν θα μπορούμε πλέον να απαγορεύσουμε τις πρακτικές που αναφέρονται εδώ. Εδώ θα μπορούσε να ισχύει κάτι τέτοιο ακόμα και για 100 εκατομμύρια ευρώ, μα κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Σχεδόν τελείωσα, παράγραφος, ε, άρθρο 28 παράγραφος 5 τώρα αναφέρομαι ε, στην ε, βοήθεια, στην αναζήτηση αποδείξεων. Εδώ προτείνεται ένας ε, κανόνας maximum από πλευρά της Κομισιόν και θα είναι πολύ δύσκολο ένας καταναλωτή να αποδείξει πως υπήρχε πραγματικά πρόβλημα εξ αρχή. Για να μπορέσει πραγματικά να τα καταφέρει θα πρέπει να έχει τεχνικές γνώσεις και θα ήταν πολύ πιο εύκολο να έχει κανείς μια διαφορετική λύση. Εδώ γίνεται επίσης λόγος για αντιστροφή του βάρους της απόδειξης και θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο ακόμα πράγματα, όπως σας το είπα και πριν από λίγο, στο επίπεδο του πεδίου εφαρμογή. Νομίζω πως ε, αν έχετε για παράδειγμα μια αγορά ε, ψηφιακών υπηρεσιών online. Τι γίνεται αν ε, κατεβάσετε ταινίες ή μουσική. Νομίζω πως αυτό που έχουμε εδώ δεν είναι κατάλληλο. Θα πρέπει και με αυτό το θέμα να ασχοληθούμε και επίσης όσον αφορά την ευθύνη του παραγωγού. Θα πρέπει, όπως ήδη αναφέρθηκε, να μιλήσουμε και για την υποχρέωση του πολιτή ή του παραγωγού απέναντι στον καταναλωτή. Εν ολίγης, ε, θα σα πω ότι η ομάδα των Πρασίνων είναι αρκετά επιφυλακτική σε σχέση με αυτά που υπάρχουν στο 4. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για λιγότερο πλήρη εναρμόνιση, εδώ μιλάμε για μικρέ βελτιώσει για ορισμένου καταναλωτές. Ελπίζω ωστόσο πω τα παραδείγματά μου έδειξαν πω τα όσα προτείνουμε εδώ μπορεί να είναι αρνητικά για εκατοντάδε εκατομμύρια ευρωπαίου καταναλωτέ. Και όπω το είπα και την τελευταία φορά κατά τη διάρκεια τη συζήτηση, εμεί. Πιστεύουμε πως θα πρέπει να γίνει κάτι για να συμβάλλουμε σε μια εσωτερική αγορά που θα λειτουργεί σωστά με υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Όμως εδώ πιστεύω πως αυτό που προτείνεται δεν είναι πραγματικά οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Γιατί η Κομισιόν λαμβάνει περισσότερο υπόψη την εσωτερική αγορά από ό,τι τον καταναλωτή. Το κεφάλαιο 4 θα πρέπει να αποσυρθεί από την οδηγία ή θα πρέπει να έχουμε ε, τελείως διαφορετικές λύσεις. Ο κύριος Βάπη μίλησε για στοχευμένη εναρμόνιση, αλλά μπορεί αυτό να είναι μια λύση, αλλά θα πρέπει να διευκρινίσει τα πράγματα, να τα ξεκαθαρίσει, γιατί δεν κατάλαβα πολύ καλά, πρέπει να σας ομολογήσω το τι εννοούσε, αλλά πάντως ε, είμαι έτοιμη να ακούσω τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι από τα διάφορα παραδείγματα που αναφέρατε καλύψατε τα τρία μεγάλα προβλήματα. Το, την εφαρμογή που είπε η κυρία Γκέφχαρτ με τους ορισμούς, πόσο θα υπάρξει εναρμόνιση, και ποιος θα υπάρχει νομική ασφάλεια και για τους καταναλωτές και για τους προμηθευτές. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπίλαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Σβάμπ για τον τρόπο με τον οποίο ε, διατύπωσε την ε, έκθεση σε συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές. Να ευχαριστήσω και τους ε, εκπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απάντησαν ευμενώς στον κύριο Σβάμπ και παρουσίασαν τις τροπολογίες στο κεφάλαιο 4, πράγμα που διευκόλυνε την εργασία μας. Θέλω να αναφερθώ σε πέντε θέματα. Καταρχήν το άρθρο 22 όσον αφορά την παράδοση όπου προβλέπεται μία προθεσμία 30 ημερών για την παράδοση ενός προϊόντος. Και εδώ συμφωνώ με τον εισηγητή ότι δεδομένη στις ε, εξελίξεως στο, ε, ε, του ηλεκτρονικού εμπορίου αυτή είναι πολύ καλή διατύπωση. Μετά το άρθρο 23 το οποίο αναφέρεται στην μεταβίβαση του κινδύνου. Πρέπει να προσπαθήσουμε να διατυπώσουμε μία διάταξη που θα λαμβάνει υπόψη ότι η μεταβίβαση του κινδύνου θα έχει άμεση σχέση με ε, την φυσική παράδοση στον καταναλωτή, διότι διαφορετικά θα προκύψουν άλλα προβλήματα σαν αυτά τα οποία σχεδιαγράφει η κυρία Γκέπχαρτ βάσει της προσωπικής της πείρας από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ένα άλλο θέμα είναι η σειρά των γεγονότων στο άρθρο 26, διότι εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο εκπροσωπώ την Πολωνία, αλλά στην Πολωνία υπάρχουν διάφορες δυνατότητες. Μπορεί ο καταναλωτής είτε να επιστρέψει το εμπόρευμα ή να το διορθώσει. Αν αυτό όμω παραμείνει στα χέρια του προμηθευτή θα μειωθούν τα δικαιώματα του καταναλωτή στην Πολωνία και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά φαινόμενα όπως παραδείγματο χάρη επανειλημμένες επισκευές ε, ε, ανικανοποιητικές ε, δηλαδή είναι μια διάταξη που θα πρέπει να εναρμονιστεί σε όλα τα κράτη-μέλη Γι' αυτό και δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένα δικαίωμα το που μπορούμε να αφαιρέσουμε από τους καταναλωτές. Μετά, η ε, καθυστέρηση ε, και η προθεσμία μέσα στην οποία ο προμηθευτής πρέπει να έχει επισκευάσει το εμπόρευμα. Δεν είναι πολύ σαφές τώρα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να το διευκρινίσουμε, διότι σήμερα μία τέτοια σάφια μπορεί να οδηγήσει σε καταχρήσεις των δικαιωμάτων κατά τρόπον ώστε να παραταθεί η περίοδος των επισκευών πέραν του εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο πρέπει να είναι αποδεκτό από τον καταναλωτή. Άρα αυτό θα πρέπει να διατυπωθεί πιο σαφώς. Ε, και τέλος ε, η περίοδος έξι μηνών η οποία προτίθεται ε, προτείνεται. Στην ε, Πολωνία έχουμε διετία, δηλαδή καλύπτουμε κατά αυτόν τον τρόπο, εξαντλούμε κατά αυτόν τον τρόπο ε, το, την περίοδο ευθύνη του πολιτή για το προϊόν που πώλησε. Ε, εάν αυτό περιληφθεί στην οδηγία ε, ε, ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα διότι παραδείγματος χάρη ε, τα καταστήματα που πουλάνε ηλεκτρικά ηλεκτρικές οικιακές συσκευές θα μπορούν να ζητούν από τον καταναλωτή να αποδείξει ότι η ζημία υπήρχε ήδη προτού παραδοθεί και παραλυφθεί το εμπόρευμα. Θα χρειαζόταν ο καταναλωτής να προσκομίσει εμπειρογνώμονες ε, με μεγάλο κόστος και αυτό θα μείωνε τα δικαιώματα των καταναλωτών και μπορεί να αποκαρδιονόντουσαν, ε, να απογοητευόντουσαν κατά αυτόν τον τρόπο οι καταναλωτές και να μην ε, ε, διεκδικούσαν τα δικαιώματά τους. Έχω επίσης και άλλες αμφιβολίες σχετικά με την εναρμόνιση της νομοθεσίας σε όλα τα κράτη-μέλη, ιδίως όταν παραδείγματος χάρη ε, τα θέματα αυτά δεν περιληφθούν διότι νομίζω ότι ε, με αυτό τον τρόπο θα μειωνόταν ε, σαφώς η προστασία του καταναλωτή. Θα αφήσω το λόγο τώρα στον κύριο Τρενταφυλλίδη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή καθώς και τους συναδέλφους που μίλησαν πριν από μένα ενεκτάσει πάνω σε ένα κεφάλαιο που ενδεχομένως να είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της οδηγίας. Θα περιοριστώ σε κάποια σημεία που αφορούν την εφαρμογή της πλήρους εναρμόνισης στο κεφάλαιο αυτό, ε, μια εισήγηση με την οποία εμείς διαφωνούμε, όπως εξάλλου και άλλοι συνάδελφοι είπαν προηγουμένως. Όπως αναφέρεται στην οδηγία, η περίοδος εγγύησης καθορίζεται στα δύο χρόνια από τη σύναψη της σύμβασης. Αυτή η ρήτρα σαφώς μειώνει το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών που ισχύει σε σειρά από κράτη-μέλη. Σύμφωνα και με την ανάλυση επιπτώσεων που έχει διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η ρύθμιση θέτει σε κίνδυνο την προστασία των καταναλωτών στις πλήστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον τα δύο χρόνια περίοδο εγγύησης αποτελούν την οροφή και συνεπώς σε πολλούς τομείς μειώνουν την περίοδο εγγύησης για τους καταναλωτές. Περιπτώσει χωρών όπου η εγγύηση επί του παρόντο είναι είτε στα πέντε χρόνια είτε και για μεγαλύτερη διάρκεια θα αντιμετωπίσουν σαφή οπισθοδρόμηση στα δικαιώματα τους από την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου. Επίση, δημιουργεί τι προποθέσει εμπορία συμβάσεων εγγύηση μεγαλύτερη των δύο ετών. Συνεπώ μια εταιρεία που πολλούσε ένα προϊόν με πέντε χρόνια εγγύηση, για παράδειγμα, θα έχει τη δυνατότητα να απολύει το ίδιο προϊόν με δύο χρόνια εγγύηση και να διαθέτει επιπλέον στη βάση του ανταγωνισμού στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς προς πώληση τη δυνατότητα αναβάθμισης της εγγύησης στα πέντε χρόνια. Άρα η μέχρι τώρα η υποχρέωση του κατασκευαστή αποτελεί πλέον προϊόν προς πώληση. Επιπλέον, η οδηγία δίνει στον έμπορο πλέον το δικαίωμα να αποφασίζει για την επιλογή των μέσων έννομης προστασίας του καταναλωτή, δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο θα αποζημιώσει τον καταναλωτή, επιδιόρθωση για παράδειγμα επιστροφή χρημάτων, αντικατάσταση προϊόντος. Μια τέτοια ρύθμιση μας βρίσκει αντίθετους γιατί στις πλήστες των περιπτώσεων ο έμπορος επιλέγει το πιο οικονομικά συμφέρον μέσο και όχι βέβαια το πιο αποδοτικό για τον καταναλωτή. Επί του συνόλου, ω πολιτική ομάδα έχουμε ενταχθεί υπέρ τη αναδιαμόρφωση του κεφαλαίου για τι εγγύησει. Η πλήρη εναρμόνιση και με το πλαίσιο το οποίο προτείνεται μα βρίσκει αντίθετου. Θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να υπάρξει μια διαφορετική ρύθμιση η οποία να αφήνει στα εθνικά νομοθετικά πλαίσια τη δυνατότητα να καθορίζουν τα ανώτατα όρια. Ταυτόχρονα να καλεί εκείνα τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν ρυθμίσει που να κατοχυρώνουν την προστασία των καταναλωτών στο πεδίο των εγγύσεων να το πράξουν ώστε να συμπεριλάβουν στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών. Για μας αγαπητοί συνάδελφοι, η προστασία των καταναλωτών αποτελεί ένα κεφαλαιόδες ζήτημα. Δεν είμαστε αρνητικοί στις προσπάθειες βελτίωσης του υφιστάμενου πλαισίου προστασίας των καταναλωτών. Αντίθετα, το επιδιώκουμε αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται με προστασία των καταναλωτών και όχι μόνο των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Πουπάκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με δεδομένο την ε, πολύ καλή δουλειά πάντα του κύριου ΣΒΑΠ αλλά και τη διάθεσή του στη συνέχεια για συνεργασία με αφορμή την εξέταση του κεφαλίου 4, παρά την αντίθεσή μου για την πλήρη εναρμόνιση σε όλα, θα ήθελα να προσθέσω κάποια σχόλια και παρατηρήσει. Ήθελα να αναφερθώ καταρχήν στο, στο άρθρο 21, αλλά συμφωνώ με τι παρατηρήσει τη κυρία Γκέπκαρτ. Στο άρθρο 22 πιστεύω ότι στι εξαποστάσεω συμβάσει, η προθεσμία παράδοση των 30 ημερών, ενώ ο καταναλωτή γνωρίζει και έχει συμφωνήσει από την πρώτη μέρα τη παραγγελία το χρόνο παράδοση, αυτό σε συνδυασμό με την έναξη της περίοδου υπαναχώρησης παρατηρώ ότι δημιουργεί κάποια αντίφαση, κάποια ανακολουθία. Τώρα, αν το εμπόρευμα δεν παραδοθεί, τότε γιατί μπορεί να μην συντρέχουν, ας το πάρουμε και έτσι, λόγια απάτης εκ μέρους του πολιτή. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αφαιθεί στην επιλογή του κατανοητή αν θα διακόψει τη σύμβαση σε περίπτωση μη παράδοση εντό 30 ημερών. Η διάταξη αυτή δεν αφορά αθέτηση συμφωνία. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, τι γίνεται σε περιπτώσεις που ο καταναλωτής ζητήσει και αποζημίωση για τυχόν βλάβη που έχει υποστεί από τη μη παράδοση εντός του χρόνου αυτού που έχουν συμφωνήσει. Ε, συνεχεία θα ήθελα να αναφερθώ στις διατάξεις του άρθρου 26, σύμφωνα με τις οποίες πιστεύω ότι μεταθέτονται οι ευθύνες του εμπόρου στον καταναλωτή, καθιστώντας τον έμπορο ανεύθυνο και τον καταναλωτή πλήρως υπεύθυνο. Συγκεκριμένα, η παράγραφος 2 σε συνδυασμό με την παράγραφο 3, στην ουσία καταργούν τα δικαιώματα υπέρ του καταναλωτή τη παραγράφου 1 που αναφέρονται και δίνουν περιθώριο επιλογή αφού τον τελικό λόγο θα έχει ο έμπορο ανάλογα με τι συμφέρει εκείνον. Δηλαδή, η παράγραφο 2 του άρθρου 26 προβλέπει ότι ο έμπορο αποκαθιστά την έλλειψη συμμόρφωση είτε με επιδιόρθωση είτε με αντικατάσταση ανάλογα με την επιλογή του. Η παράγραφο 3 προβλέπει ότι αν ο έμπορο έχει αποδείξει ότι η αποκατάσταση έλλειψη υπομόρφωση με επιδιόρθωση αντικατάσταση είναι παράνομη, αδύνατη ή θα προξενούσε τον έμπορο δυσανάλογη προσπάθεια, τότε μόνο ο καταναλωτή μπορεί να επιλέξει τη μείωση τη τιμή ή την κατάργηση τη σύμβαση. Εμά στην ελληνική νομοθεσία, σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντο, ο καταναλωτή μπορεί να επιλέξει ή τη διόρθωση, ή την αντικατάσταση, ή τη μείωση τιμή, ή την αναστροφή τη πόλη ο ίδιο καταναλωτή. Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο 26, στην παράγραφο 4β, Προβλέπετε ότι ο καταναλωτή μπορεί να επιλέξει μία από τι τέσσερι μορφέ αποκατάσταση όταν ο έμπορο δεν προβεί στην αποκατάσταση τη έλλειψη συμμόρφωση εντό ευλόγου χρονικού διαστήματο ή η ίδια βλάβη επανεμφανίστηκε περισσότερο από μία φορά εντό μικρή χρονική περίοδου. Δεν θα πρέπει να οριστεί ποια είναι η διάρκεια του εύλογου χρονικού διαστήματο ή ποια η διάρκεια τη μικρή περίοδου. Τέλο, αναφορικά με τι εμπορικέ εγγυήσει, θα ήθελα να προσθέσω ότι ίσω θα πρέπει να εξεταστούν αν μπορούν να μεταβιβαστούν σε επακόλουθο αγοραστή αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε γιατί ένα καταναλωτή να αγοράσει ένα ελαφρώ μεταχειρισμένο προϊόν, αν δεν έχει κάποια εγγύηση. Ευχαριστώ πολύ. λοιπόν, πριν δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή, υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις εκ μέρους των μελών. Όχι. Ωραία λοιπόν, μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις θα δώσω το λόγο και έχετε πολύ χρόνο στη διόθεσή σας ε, στην Επιτροπή, στον κύριο Τζοτζέπε Μόντι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και καλησπέρα σας όλοι. Έχω να απαντήσω πολλές ερωτήσεις. Ελπίζω λοιπόν ότι μπορώ να υπολογίσω στα θετικά σας συναισθήματα και στην ανοχή σας για να είναι οι απαντήσεις μου αρκετά ξεκάθαρες. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι κατάλαβα τα πρώτα σχόλια του Ανδρέα Σβάμπ ότι δεν έχει ακόμα μια ξεκάθαρη εικόνα της οδηγίας, γιατί είναι εξαιρετικά πολύπλοκο νομοθέτημα, το οποίο συγχωνεύει τέσσερις υπάρχουσες οδηγίες και ε, περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η σχέση μεταξύ των δικαιωμάτων των καταναλωτών έτσι όπως αναφέρονται στην οδηγία και τα συμβατικά δίκαια στις χώρες μέλη δεν είναι πάντοτε απολύτως ξεκάθαρα. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εργαζόμαστε πολύ σκληρά στο Συμβούλιο ούτε ώστε να διασφαλίσουμε ότι ενδεχομένως θα υπάρξει μια σαφήνεια στο κείμενο όσον αφορά τα δικαιώματα που προβλέπονται από την οδηγία και συγκεκριμένα ε, και, και, τα, τις συμβατικές ε, υποχρεώσεις, το δίκαιο των συμβατικών υποχρεώσεων. Τώρα, η λογική πίσω από την πρόταση της ε, πλήρους αναρμόνησης θέλει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ε, καταναλωτών και των εμπόρων στην εσωτερική αγορά. Δεν συμφωνούμε με την κυρία Τουλούμεν ότι τα συμφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρηματιών είναι ανταγωνιστικά. Αν οι καταναλωτές δεν έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν από έναν έμπορο που βρίσκεται σε μια άλλη χώρα μέλος, αυτό σίγουρα δεν είναι ισόφελος του καταναλωτή. Ή εάν ο καταναλωτής δεν έχει πρόσβαση σε ανταγωνιστικές προσφορές, ε, ε, μειώνονται τα ωφέλη. Η κατάτμιση των, ε, των δικαιωμάτων του καταναλωτού και ο συνδυασμός με τις ε, εθνικές διατάξεις δημιουργεί σημαντικούς φραγμούς για την εσωτερική αγορά. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι έμποροι αποφασίζουν να μην πωλήσουν σε καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι σε άλλη χώρα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αλλάξει αυτή η κατάσταση, γιατί εκεί όπου το δικαστήριο αποφάσισε μια εταιρεία που έχει μια ιστοσελίδα και είναι προσετή από τους καταναλωτές στο εξωτερικό, απευθύνει τις δραστηριότητές της προς ε, καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό, όλοι οι φόβοι και ενισχύσεις των εμπόρων, ίσως εάν ε, εμπλακούν σε μια διασυνοριακή συναλλαγή, και τελικά ε, συρθούν ενώπιον του δικαστηρίου του, της χώρας του καταναλωτού, επικυρώνονται αυτοί οι φόβοι. Θα ήθελα να πω ορισμένα ε, λόγια για την πλήρη εναρμόνιση όταν κάνουμε την αξιολόγηση των επιπτώσεων, η πλήρη εναρμόνιση ήταν μία από τι δυνότητε που εξετάσαμε. Εξετάσαμε επίση τη δυνατότητα, γιατί θέλαμε πραγματικά να ολοκληρώσουμε την ιστορική αγορά σε αυτό το τομέα. Αυτό ήταν ο στόχο τη μεταρρύθμιση. Μία από τι δυνατότητε τη πολιτική ήταν πλήρη εναρμόνιση και είχαμε την αίσθηση ότι η πλήρη εναρμόνιση ήταν ο μόνο τρόπο για να, επιτυχάνουμε τους ζητούς να επιτύχουμε συγγνώμη, του ζητού στόχου τη μεταρρύθμιση. Δηλαδή να δημιουργήσουμε μια, ένα πιο προβλέψιμο ρυθμιστικό ασφαλιστικό περιβάλλον τόσο για τον επιχειρηματή όσο και για τον καταναλωτή. Και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να μπούμε σε μια συζήτηση ε, περί των αρχών, ε, θεωρητική, για την πλήρη εναρμόνιση σε αυτή τη φάση. Γιατί επιλέξαμε να μην το κάναμε στο Συμβούλιο, στην ομάδα εργασία, στο Συμβούλιο. Πραγματικά προσπαθήσαμε να είμαστε ρεαλιστέ, πραγματιστέ. Ε, δηλαδή, ανατρέχουμε τι διατάξει τη οδηγία μία προ μία και μόνο εφόσον έχουμε διευκρινίσει τι προθέσει τη Επιτροπή και έχουμε ε, αποφασίσει για το περιεχόμενο των διατάξεων, ε, μπορεί τότε να αρχίσουμε τη συζήτηση για το επίπεδο εναρμόνησης. Δυστυχώς ο εισηγητής έφυγε γιατί ήθελα πραγματικά να απαντήσω τις ερωτήσεις του. Παρ' όλα αυτά θα το κάνω έμεσα. Επιτρέψατε μου να πω κάποια πράγματα το κεφάλαιο 4 πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ των άρθρων 22 και 23 τα οποία είναι ολοκένουργια. Ε, επιστρέφει ο εισηγητής το 22 και το 23 που είναι νέα και τα οποία ε, τόνισε ο κύριος, όπως τόνισε ο κύριος Βέλλον αφορούν ε, σημαντικά θέματα στην οικονομία δηλαδή την παράδοση και τη μεταβίβαση του κινδύνου. Σε αυτές οι διατάξεις εθετήσαμε μία προσέγγιση ιδιαίτερως φιλική προς τον ε, καταναλωτή. Απαντώ την ερώτηση της κυρίας Σβάμπ. Ποιος είναι υπεύθυνο εάν απολεσθούν τα είδη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Είναι ο έμπορος ο οποίος είναι υπεύθυνο. Είναι πώς ο καταναλωτής ε, προστατεύεται έως ότου αποκτήσει την φυσική κυριότητα του αγαθού, του είδους και με καταπλήσει το ότι η κυρία Γκέπαρτ δεν το τόνισε, γιατί θα έπρεπε να δηλώσει ότι είναι ικανοποιημένη από αυτό το αυξημένο επίπεδο προστασίας του καταναλωτού. Δεν το έκανε όμως. Τώρα, η διάρκεια της εγγύησης και το βάρος της απόδειξης. Εδώ, η διάκριση μεταξύ ε, νέων άρθρων του 22 και του 23 και των άλλων άρθρων τα άλλα άρθρα δεν είναι νέα άρθρα, δεν είναι νέα δικαιώματα. Αυτό που κάναμε είναι να ε, δούμε ήδη τις υπάρχουσες διατάξεις, να βελτιώσουμε την γλωσσική τους διατύπωση στα αγγλικά, αποφύγαμε τη διπλή άρνηση, ε, προσπαθήσαμε να εθετήσουμε ένα πιο κομψό ύφος στην πρόταση, γλωσσικό ύφος και αναφερθήκαμε στα υφιστάμενα δικαιώματα των καταναλωτών. Δηλαδή, πολλά από τα ερωτήματα της κυρίας Κέπερ αφορούν την υπάρχουσα οδηγία του 99. Όλες οι ερωτήσεις για το άρθρο 24, γάμα, για το 23, για το 24, παράγραφος 3, δεν είναι νέα δικαιώματα, δεν είναι νέοι κανόνες, είναι τα υπάρχοντα δικαιώματα τα οποία ε, ε, διατυπώνονται στην ε, παλαιά οδηγία του 99. Θα σας απαντήσω όμως στις ερωτήσεις σας. Είναι αλήθεια ότι ακολουθήσαμε την προσέγγιση της πλήρους εναρμόνισης και επιλέξαμε αυτό το οποίο επιθυμούμε. Θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ενδεδειγμένο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις διατυπώσαμε τις ελάχιστε προδιαγραφέ και τις μετατρέψαμε σε πλήρη εναρμόνιση, γιατί θεωρήσαμε ότι πλήρη εναρμόνιση ε, που προβλέπει η ισχύουσα οδηγία ήταν επαρκή. Θα πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά τι ανησυχίε των καταναλωτών, η αρχική μας εντύπωση επικυρώθηκε από μια έρευνα για την συμπεριφορά και τις στάσεις των καταναλωτών όσον αφορά ε, τα μέσα διόρθωσης ή παρέμβαση σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων. Ε, υπάρχει λοιπόν αυτή η παρεμβαση σε περιπτωση ελαττωματικων προιοντων υπαρχει λοιπον αυτη η ερευνα Θα ήθελα πραγματικά να σας παρουσιάσω τα ευρήματα ή τα συμπεράσματα στο εγγύς ε, μέλλον στην Επιτροπή σας. Ένα θέμα το οποίο τέθηκε μεταξύ άλλων από την κυρία Τορούνεν ε, των ε, μέτρων υπέρ των ε, καταναλωτών και των παραδοσιακών τρόπων παρέμβασης στις χώρες μέλη. Νομίζω θα πρέπει πράγματι να υπάρχει μεγαλύτερη καθαρότητα στο κείμενο. Γιατί τώρα όλοι αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση αοριστίας. Ε, Συμφωνώ ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο αυτή η σχέση. Η πρόθεσή μας, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν να επηρεάσουμε την ελευθερία των χωρών μελών να ε, παραμείνουν στα παραδοσιακά τους ε, συμβατικά μέτρα τα στην Ιταλία και λοιπά ή τις εγγύσεις που προβλέπονται στη Γαλλία από το γαλλικό σύστημα. Στο Συμβούλιο προσπαθούμε να κάνουμε μια πολύ προσεκτική δουλειά και βλέπουμε σε ποια έκταση η προστασία των καταναλωτών, δηλαδή κατά πόσο μπορούμε να πάμε πιο μακριά στην εναρμόνιση των δικαιωμάτων, εισάγοντας για παράδειγμα ένα δικαίωμα απόρριψης το λεγόμενο right to reject, ε, παρόμοια με αυτό που υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία ή να καθισχάσουμε τους φόβους της Γαλλίας ε, προεκτείνοντας τη διάρκεια της εγγύησης ή βρίσκοντας κάποια άλλη λύση στο ζήτημα της εγγύησης. Ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό και που θα ήθελα να τονίσω αφορά το κεφάλαιο 4 σε σχέση με τα είδη, το οποίο αφορά τα είδη, τα προϊόντα και όχι τις υπηρεσίες. Δεν αφορά τις υπηρεσίες, γιατί καμιά φορά οι λύσεις που βλέπετε το κεφάλαιο 4 δεν ε, αφορούν τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, κυρία Τερούν, αν πάτε στον κομωτή και σας κόψει άσχημα τα μαλλιά σας, ασφαλώς δεν θα ζητήσετε μία αντικατάσταση, μία επιδιόρθωση. Ε, και αυτό είναι το θέμα που ήθελα να θίξω δεν είναι κάτι το οποίο ρυθμίζεται στην οδηγία αυτή. Είναι κάτι που είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής αυτής της οδηγίας ή της εμβέλειας αυτής της οδηγίας και θα συνεχίσουμε τη ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο στην περίπτωση αυτή. Το ίδιο ισχύει και για τις ε, ψηφιακές υπηρεσίες. Το κεφάλαιο 4 αφορά μόνο αυτά υλικά αγαθά, ενώ τα ψηφιακά δεν είναι, είναι και οι υπηρεσίες στην περίπτωση αυτή αφορούν τις εκχωρήσεις ε, αδειών ε, ε, πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ. Και το πεδίο αυτό θα συνεχίσει να ρυθμίσει σε εθνικό επίπεδο. Εμείς ήδη ξεκινήσαμε ένα πολύ, πολύ μακρόπρονες έρευνες για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές online σε σχέση με τα εθνικά δίκαια όσον αφορά αυτές τα, τα, τις ψηφιακές υπηρεσίες. Είναι η έρευνα που αφορά τα ψηφιακά προϊόντα σε συνάρτηση με τα ισχύοντα δίκαια ε, στις χώρες μέλη. Um, Uh, I think was Mr. Poupakis. Uh, I... Νομίζω ο κύριος Πουπάκης, ε, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, ανέφερε το θέμα της ατελούς εναρμόνισης του κεφαλαίου 4. Όταν λέει για παράδειγμα ότι δεν ρυθμίζουμε το δικαίωμα για βλάβες, ε, και πάλι αυτό που κάναμε εδώ δεν είναι ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, δεν είναι ένα ευρωπαϊκός ε, αστικός κώδικας. Έχουμε ακολουθήσει αυτό που λέμε full targeted harmonization, δηλαδή πλήρως στοχοθετημένη εναρμόνιση. Έχουμε επιλέξει μερικά συγκεκριμένα ε, θέματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά σε διασυνοριακές συναλλαγές και, και επιλέξαμε να τα εναρμονίσουμε πλήρως, έτσι ώστε να υπάρχει... Ε, αλληλεπίδραση με τις διατάξεις του αστικού κώδικα στα κράτη-μέλη. Και έτσι λοιπόν, αν καταναλωτή ε, υποστεί βλάβη λόγω καθυστερημένης παράδοσης ή λόγω μη παράδοσης, η οδηγία δεν δεν ε, αναιρεί το δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει αποζημίωση από τον έμπορο. Τέλος. Νομίζω ότι ολοκλήρωσα και ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις της κυρίας Γκέμπχαρτ. Σύμφωνο, γιατί έλεγα να σας πω ότι δεν απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Στο, στο άρθρο 22 παράγραφος 2. Ποια είναι η περίοδος παράδοσης. Η περίοδος παράδοσης είναι η περίοδος που συμφωνείται από τα μέρη στην περίπτωση έλλειψης συμφωνίας είναι 30 μέρες. Και έπειτα ο κανόνας, ε, η ρύθμιση είναι πολύ υδρακόντια. Είναι υπέρ του καταναλωτή. Αν ο έμπορος δεν μπορέσει να ε, τηρήσει τη σύμβαση, τότε ο καταναλωτής μπορεί να καταργήσει τη σύμβαση και να ζητήσει πίσω τα χρήματά του. Αυτό σημαίνει ότι είτε θα πρέπει να επιμείνει για την εκτέλεση της σύμβασης, είτε μπορεί να ζητήσει αποζημιώσεις. Έπειτα, το παράδειγμα της μεταφοράς της πραγματικής κατοχής του αγαθού. Τι συμβαίνει δηλαδή αν ο έμπορος, για παράδειγμα, δώσει το αγαθό σε κάποιο γείτονα, παραδώσει το αγαθό σε κάποιο γείτονα ή που, που, παριστάνει ότι είναι ο γείτονας και ο οποίο εξαφανίζεται με το του αγαθού. Εκεί ε, έχουμε μία ε, αμελή εκτέλεση της σύμβασης, γιατί η διάταξη είναι σαφής, ότι δηλαδή τα, αγαθά θα πρέπει να παραδοθούν στον καταναλωτή είτε σε κάποιον άνθρωπο που ορίζει, που ορίζει ο ίδιος ο καταναλωτής. Όχι σε οποιοδήποτε γείτονα, το οποίο το όνομα δεν έχει ποτέ αναφερθεί από τον ίδιο τον καταναλωτή. Άρθρο 24, παράγραφος 3. Um, in which situations... Uh, Σε ποιες περιπτώσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορέσει να ζητήσει αποκατάσταση. Το 24-3. Ωραία. Λοιπόν, σε ποιες περιπτώσεις ο καταναλωτής γνώριζε ή έπρεπε να γνώριζε το ελάττωμα. Ας πούμε, πες ότι, πείτε ότι πας σε ένα κατάστημα επίπλων και ότι υπάρχει ένα ε, αντικείμενο το οποίο είναι γρατζουνισμένο και φαίνεται και άρα ο καταναλωτής παίρνει και μια έκπτωση 20% ας πούμε λιγότερο για, το, για ένα τραπέζι λόγω αυτής της γρατζουνιάς. Άρα λοιπόν εκεί ο καταναλωτής δεν μπορεί να ζητήσει αποζημίωση αφού γνώριζε το ελάττωμα. Ήταν εμφανές. Αυτό δεν είναι τίποτα νέο. Αυτό ήδη υπάρχει στην ε, οδηγία για τις πωλήσει. Άρθρο 24.4c, όπου λέει ότι ο έμπορος δεν θα δεσμεύεται από δημόσιες δηλώσεις για παράδειγμα, αν η απόφαση να αγοράσει κανείς τα αγαθά δεν μπορούσε να επηρεαστεί, αν η απόφαση του καταναλωτή να αγοράσει τα αγαθά δεν μπορούσε να επηρεαστεί από τη δήλωσή του και πάλι δεν είναι τίποτα νέο, εδώ έχουμε αντιγράψει την ισχύουσα διάταξη, αλλά τι σημαίνει. Σημαίνει πως αν ο καταναλωτής ε, έχει μπροστά του μια υπερβολική δήλωση, ας πούμε ότι συναντά τους ωραιότερους ανθρώπους, του, τους καλύτερους ανθρώπους στον κόσμο αν οδηγεί το γιώτα, αυτοκίνητο το αυτό δεν ε, θα το πάρει σοβαρά κανένα καταναλωτή και ακριβώς αυτό το θέμα είναι που ρυθμίζεται εδώ σε αυτή τη διάταξη. The, um, the, provision uh... I mean, the, the, good question asked by, by, by Mrs. Gephardt concerning uh, the compatibility between the είπε η κυρία Γκέπχαρτ τώρα για τη συμβατότητα ανάμεσα στην εμπορική εγγύηση και το γεγονός ότι ο καταναλωτή θα πρέπει να είναι ενήμερος, να ενημερώνεται μάλλον όταν χρειάζεται να μεταφέρει την εμπορική εγγύηση στον επόμενο αγοραστή και τη διάταξη στο γκρι, στο, στο, στην γκρίζα λίστα που εμποδίζει τους εμπόρους να το καταστήσουν δυσκολότερο για τους καταναλωτές που μεταφέρουν τα αγαθά. Για παράδειγμα, μάλλον συμπεριλαμβανομένη της μη με, δυνατότητας μεταφοράς της εγγύησης. Υπάρχει μια γκρι λίστα, δηλαδή μια θεώρηση αδικίας που μπορεί να την αντικρούσει ο έμπορος. Αλλά μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις όπου να είναι απόλυτα θεμητό ένας έμπορος να προσπαθήσει να περιορίσει τη δυνατότητα μεταφοράς της εμπορικής εγγύησης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα ένα μικρό, μια μικρή βιοτεχνία ενό ανθρώπου στη Νότια Ιταλία που παράγει. Εγώ έρχομαι από τη Νότια Ιταλία που φτιάχνει, α πούμε, μαντολάτο. Ένα τέτοιο άνθρωπο μπορεί να δίνει μια εμπορική εγγύηση που περιορίζεται στα δύο χρόνια, αλλά που περιορίζεται στους ανθρώπους που κατοικούν εκεί. Γιατί θα ήταν εξαιρετικά βαρύ να ε, ε, εγγυηθεί σε έναν αγοραστή που πάει να ζήσει στο, που ζει στο Όσλο ή στη Σκοτία. Μπορεί να υπάρχουν ε, περιπτώσεις δηλαδή όπου για τον πολιτή είναι απαραίτητο να περιορίσει τη γεωγραφική το γεωγραφικό, τη γεωγραφική ισχύ της εγγύησης. Νομίζω πως ήδη απάντησα σε περισσότερες ερωτήσεις, αν όχι σε όλες. Διαφορετικά, Είμαι στη διάθεσή σας. Euh, Ευχαριστώ. Να σα φέρω εγώ, να σας δώσω κι εγώ μια δική μου σκέψη. Νομίζω πως γίνεται όλο και πιο περίπλοκο το πράγμα. Να το λέω επειδή είμαι πρόεδρος και έχω το λόγο, έτσι κι αλλιώς αλλά τα δικαιώματα του καταναλωτή είναι κάτι τα οποία θα πρέπει εμείς να τα συντάξουμε με σε ξεκάθαρο τρόπο. Ευανάγνωσταν, αλλά δεν πειράζει, δύσκολα ξεκινάμε, αλλά μόλις ξεκινάμε, οπότε θα τα απλοποιήσουμε. Ίσως να μπορούσαμε να έχουμε ένα άλλο φως, θα αφήσω το λόγο στην Σουηδική Προεδρία, στον κύριο Άντρες Δελίνς, ο οποίος πιστεύω έχει συμμετάσχει σε πολλές συνεδριάσεις. Eh, jag kan kort redogöra för arbetet i rådet under hösten. Vi har hållit ett eh, större antal arbetsmöten och arbete... Ναι, έχω που έγιναν το Έχουμε λοιπόν ε, κείμενα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί πλήρως ε, στο Συμβούλιο. Είμαστε στο κεφάλαιο 2 και αύριο έχουμε το Συμβούλιο περί και αύριο το απόγευμα θα συζητήσουμε τα θέματα καταναλωτή και οι υπουργοί των διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν ήδη προετοιμαστεί για να οργανώσουμε την αυριανή συζήτηση και έχουμε συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν ε, το κεφάλαιο 3, όπως η εξαποστάσεως πωλήσει, η διαλογραφίας πωλήσει και έχουμε και κάποιες γενικές ερωτήσεις για το κεφάλαιο 4 που εξετάστηκε σήμερα και έχουμε και σημαντικά θέματα για το πεδίο εφαρμογή και το κατά πόσο ή σε ποιο βαθμό η οδηγία αυτή θα πρέπει να καλύπτει και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Και έχουμε την πρόθεση να κάνουμε αυτή τη γενική συζήτηση για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε κάπως την εικόνα, να βρούμε κάποιους προσανατολισμούς από το Συμβούλιο των Υπουργών. Από την άποψη της Σουηδίας και της Σουηδικής ε, Αντιπροσωπείας, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πω ήταν εξαιρετικά επικοδομητικά κατά τη διάρκεια της συζήτησης και η συζήτηση αυτή θα μας επιτρέψει να δούμε πιο ξεκάθαρα τα πράγματα για τις μελλοντικές μας συζητήσεις. Και κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων η Σουηδική Προεδρία κάνει μια γενική ανακεφαλαίωση των όσων κάναμε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στο πλαίσιο αυτού του εγγράφου θα ξαναδούμε τα διάφορα κεφάλαια της πρότασης. και οι Υπουργοί Αρμόδιοι περί κατανάλωσης έχουν αναλάβει να συζητήσουν το θέμα στις 17 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Όλα είχαν προετοιμαστεί, αλλά από ό,τι καταλάβαμε μετά από μια αλλαγή του χρονοδιαγράμματος δεν θα καταστεί δυνατό να έχουμε τη συνεδρίαση αυτή στο Στρασβούργο στις 17. Πραγματικά λυπούμεθα πολύ, αλλά Εν πάση περιπτώσει, η Σουηδική Προεδρία είναι στη διάθεσή σας αν έχετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Merci Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Υπογραμμίσατε όντως δύο σημαντικά προβλήματα. Στις πολλές εξαποστάσεις και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ο κύριος Άντριου ο κύριο Χάρμπορ θέλει να διευκρινίσει κάτι. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήθελα σύντομα να απαντήσω στα όσα είπε το Συμβούλιο για τη συνεδρίαση τη 17 η και ίσω και να καταγραφεί στα πρακτικά το γεγονό ότι είμαστε ιδιαίτεροι Ιδιαίτερα ευγνώμονε στην Υπουργό που ήθελε να έρθει να μα ενημερώσει για την πρόοδο, για την οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Όπω γνωρίζετε, προγραμματίζαμε να γίνει αυτό, αλλά δυστυχώ η Προεδρία τώρα έχει βάλει δύο προφορικές ερωτήσεις για την, για την Επιτροπή μας, για την Πέμπτο πρωί. Δυστυχώς δεν ε, την κάνουμε εμείς την ημερήσια διάταξη και για την ώρα αυτή παραμένει η θέση. Έτσι έχουν τα πράγματα προς λύπη μου. Πραγματικά θα πρέπει να διαβιβάσετε τη λύπη μας στην κυρία Σαμπούνη. Δεν είναι που δεν θέλουμε να την ακούσουμε, αλλά δυστυχώς το χρονοδιάγραμμα στο Στρασβούργο δεν μας επιτρέπει να οργανώσουμε και άλλη συνεδρίαση για την Πέμπτη. Επίσης θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη, προσπαθήσαμε μάλλον να οργανώσουμε τηλεδιάσκεψη, ούτε γι' αυτό είχαμε χρόνο. Θα βρούμε κάποιον άλλο τρόπο να επικοινωνήσουμε, γιατί πιστεύω πως όλοι μας είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Γιατί ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η επίσκεψη που είχαμε και τον ε, Σεπτέμβριο. Επίσης να πω πως και η κυρία Μπούλινγκ ήθελε να συναντηθούμε, αλλά δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα όταν προσπαθούμε να τα στριμώξουμε όλα στο τέλος κάθε προεδρίας. Ωραία, μας μένει ακόμα χρόνος. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Τούρινεν, στην κυρία Γκέπχαρτ και τέλος τον κύριο Σβάμπ, τον κύριο Συγγητή, η Μαντάμ Τούρινγκεν. Ναι, θα είμαι πολύ σύντομη. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο μόλις είπε η Επιτροπή. Είπατε ότι υπάρχει μια νέα εκδοχή τώρα. Ε, είπατε ότι δεν υπάρχουν μεν πάρα πολλές αλλαγές, αλλά όταν πηγαίνουμε από ένα ελάχιστο στις, σε όλες τις διατάξεις, αυτό συνεπάγεται πάρα πολλές αλλαγές για πολλούς ανθρώπους και θα πρέπει κανείς να τοποθετηθεί έναντι αυτής της κατάστασης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τα ίδια όπως προηγουμένως. Ορισμένες χώρες σήμερα έχουν καλύτερες ρυθμίσεις από αυτό το οποίο προβλέπετε εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω και πάλι να σας ζητήσω μάλλον να εξηγήσετε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι τα πράγματα παρέμειναν τα ίδια και αυτό είναι εις τους. Οι Εθνικές Οργανώσεις Καταναλωτών και οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις Καταναλωτών, οι Σύλλογοι Καταναλωτών ε, είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Δεν, γνωρίζουν, δεν αναγνωρίζουν αυτά τα πλεονεκτήματα της νέας ρύθμισης. Εγώ δεν είμαι κατά της εναρμόνισης. Το θέμα είναι ε, πιο γνώμονα θα πρέπει να ακολουθήσουμε και πού θα πρέπει να βάλουμε τον πύχη. Κατά τη γνώμη μου, ο πύχης είναι πολύ χαμηλά. Γιατί δεν βάζουμε τον πύχη λίγο ψηλότερα, γιατί εάν το κάνουμε μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό καλά και στους καταναλωτές. Ε, αναφερθήκατε σε διασυνοριακά ζητήματα αλλά ακριβώς αυτές οι ψηφιακές υπηρεσίες, δηλαδή η μουσική στο ίντερνετ, το να την αγοράζει και να την κατεβάζει από το ίντερνετ, αυτό είναι ιδιαίτερο διασυνοριακό και αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, ιδίω τη γενιά μου και θα έχει όλο και σπουδάτερη θέση στο μέλλον. Συνεπώ θα πρέπει να σκεφτούμε και ε, αυτό ως διασυνοριακό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκέπχαρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση θα πρέπει να πω όπου πάντοτε ε, όπου μεγαλώνουν και διαβεβαιώσει, αυξάνονται μάλλον οι διαβεβαιώσει και από την ε, Επιτροπή ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά πολύπλοκο ζήτημα έχω την εντύπωση ότι δεν καταλαβαίνουμε απολύτως περί τίνος πρόκειται. Θα πρέπει να το θέσουμε έτσι. Και αυτό δεν το εννοώ τώρα προσωπικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα, ε, να αναφερθούμε ξεκάθαρα στην επιχειρηματολογία. Είπατε, ναι μεν, ισχύει αυτό, αλλά τα κείμενα είναι τα ίδια. Και τα σημεία κριτικής που διατύπωσα ε, αφορούν το παλαιό κείμενο. Αλλά εγώ διατύπωσα αυτή την κριτική και στο παρελθόν. Φυσικά τα κείμενα μοιάζουν μεταξύ τους, εκτός από το άρθρο 26 όπου υπάρχει μια ξεκάθαρη επιδείνωση των δικαιωμάτων καταναλωτών. Θα πρέπει να το πούμε ρητά, γιατί στο αρχικό κείμενο ο καταναλωτής είχε το δικαίωμα επιλογής, κάτι το οποίο πλέον είναι εντελώς αδύνατο. Το δικαίωμα επιλογής ε, παραχωρείται αποκλειστικά στου πολιτέ. Και αυτή είναι μια ξεκάθαρη επιδείνωση έναντι του αρχικού κειμένου. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Συγκρίνεται δύο ευρωπαϊκά κείμενα. Το ένα είναι πλήρως εναρμονισμένο, το άλλο είναι εναρμονισμένο σε ένα ελάχιστο επίπεδο. Και αυτή τη διάκριση θα πρέπει να την έχετε κατά νου, ότι στις χώρες μέλη υπάρχουν πολλές ε, διαφορές όσον αφορά το ισχύον δίκαιο. Και ε, από αυτό το ίδιο κείμενο, εκεί που είναι περίπου το ίδιο, όπως είπατε, ε, στις χώρες ε, μέλη αυτό συνεπάγεται μία μείωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Και εμείς δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Δεν επιθυμούμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο ως μέλη της Ευρωβουλής. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Ε, δεν, δεν είστε εσείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα πρέπει να ε, σταθείτε υπόλογοι εναντί των πολιτών. Εμείς είμαστε υπόλογοι εναντί των πολιτών, εμείς είμαστε οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών που πρέπει να τους εξηγήσουμε τι κάνουμε ακριβώς στο ευρωπαϊκό πλαίσιο όσον αφορά την νομοθεσία. Ναι, το να πούμε δεν έχετε πλέον το δικαίωμα ή έχει μειωθεί το διάστημα της εγγύησης ή σε ορισμένες περιπτώσεις παρατείνεται, αλλά η χρονική στιγμή ε, που υπολογίζει κανείς τοποθετείται νωρίτερα κλπ. Άρα συνεπώς πράγματι η διάρκεια αυτή μειώνεται. Ε, πώς θα πρέπει να τα εξηγήσει κανείς όλα αυτά στους πολίτες και να πει ε, ότι απλουστεύοντας το κείμενο αυτό, παρόλο που δεν νομίζω ότι προκύπτει από τη συζήτηση ότι πράγματι το απλουστεύσαμε, προχωράμε σε μια εναρμόνιση γιατί τελικά να είναι όλοι σε ίση κατάσταση, αλλά να συρκρώνονται τα δικαιώματά τους, να επιδεινώνεται η κατάσταση των καταναλωτών. Νομίζω γι' αυτό θα πρέπει να συζητάμε. Ε, δεν πρόκειται για τη σύγκριση του κειμένου όπως ήταν πριν και όσα έχει σήμερα, αλλά σε σύγκριση με αυτό που γίνεται στο επίπεδο των χωρών μελών. Αυτό είναι ο γνώμονας της σύγκρισης και αυτό παραβλέπεται συστηματικά, φοβούμε στη συζήτηση, στην τρέχουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κέπαρτ. Νομίζω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις σήμερα στην εσωτερική αγορά για το θέμα αυτό φτάνουν σε ένα σημείο για το Συμβούλιο όπου η Σουηδική Προεδρία ε, συνειδητοποιεί την ε, πολυπλοκότητα αλλά και το ζήλο που έχουμε ως προς το θέμα αυτό. Ε, κύριε Σβάμπ, θέλετε να πάρετε το λόγο ή με επιτρέπετε προηγουμένως να δώσω για λίγα λεπτά στην Επιτροπή εάν θέλει να απαντήσει για να διευκρινίσει λίγο τη θέση της. Ε, η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Οι απαντήσεις είναι πολύπλοκες γιατί οι ερωτήσεις είναι πολύπλοκες ώρες οι ερωτήσεις που έθεσε η κυρία Κέπαρτ είναι βεβαίω θεμητέ, αλλά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκε. Και ε, συνεπάγονται περίπλοκες απαντήσει. Είναι πολύπλοκο το ζήτημα. Ρυθμίζουμε ένα, μια σειρά θεμάτων που κατέχουν μια θέση κλειδί όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Και η κυρία Τουρούρερ και η κυρία Κέπχερτ πάντοτε επιμένουν σε επίπεδο προστασίας. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ναι μεν το επίπεδο προστασία είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πιστεύουμε ότι η οδηγία ως έχει αυτή τη στιγμή βασίζεται ή μάλλον επιτυχάνει ένα υψηλό, ένα υψηλό κοινό επίπεδο προστασίας και η πλήρης εναρμόνιση την οποία, στην οποία αποβλέπει η οδηγία θα καταργήσει κάποιους φραγμούς της εσωτερικής αγοράς και από αυτή την κατάργηση θα επωφεληθούν οι καταναλωτές, γιατί θα έχουν περισσότερες διασυνοριακές προσφορές. Ε, λόγω αυτών των ρυθμιστικών ε, φραγμών, οι καταναλωτές είναι εγκλωβισμένοι ε, εντός αναθερικών συνόρων. Όταν ε, ε, ασχοληθήκαμε με το θέμα του, των πωλήσεων εξ υπήρχε ένας αρχικός ο οποίος μου έλεγε πάντοτε ότι το θέμα αυτό είναι νομικά ιδιαίτερος ε, πολύπλοκο, διότι υπάρχει ακριβώς κατάτμιση των νομικών συστημάτων. Γιατί να μπω στον κόπο να πωλήσω σε έναν ε, καταναλωτή στην Κύπρο, ε, παρόλο που υπάρχουν κοινά, υπάρχει ένα κοινό δίκαιο, ή στη Μάλτα. Συνεπώς, ο πραγματικός κίνδυνος, εάν δεν εναρμονίσουμε αυτούς τους κανόνες, είναι ότι οι καταναλωτές στις περισσότερες χώρες θα ε, ε, ε, εξοβαλιστούν από την εσωτερική αγορά. Οι ψηφιακές υπηρεσίες, τα όσα είπε η κυρία Τορούνεν, πιστεύω ότι η οδηγία, βεβαίως υπάρχουν κάποιες διατάξεις όπως είναι το κεφάλαιο 5 στην οδηγία, που αναφέρονται πλήρως στις ψηφιακές υπηρεσίες η, παράδειγμα, οι διατάξεις για τις εξαποστάσεις συμβάσεις αφορούν εν μέρη τις ψηφιακές υπηρεσίες. Νομίζω ότι ασχολούμεθα εδώ με ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά πολύπλοκο. Εάν θέλουμε να περιλάβουμε και τις ψηφιακές υπηρεσίες, για παράδειγμα να παρατείνουμε ε, την προστασία εκεί, να επεκτείνουμε την προστασία εκεί, νομίζω ότι θα ασχολούμαι με κάτι το οποίο είναι εντελώ πολύπλοκο και το οποίο πλέον δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε. Παρ' όλα αυτά, συμμερίζομαι την άποψή σα ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να αναλύουμε τα προβλήματα που αφορούν τι ψηφιακέ υπηρεσίε. Θα το κάνουμε ε, και πραγματικά ε, θα δώσουμε πολλά χρήματα προ αυτή την κατεύθυνση και θα δούμε τι θα βγει από αυτέ τι έρευνε. Θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών μαζί σα. Τέλο, το θέμα ε, τη κυρία Κέπχαρτ όσον αφορά το άρθρο 26 και τη δυνατότητα επιλογή. Ποια είναι η κατάσταση, κατά την άποψή μου, εάν ε, θέλετε να είμαι 100% ειλικρινής μαζί σας, τίποτα δεν αλλάζει. Τώρα ο καταναλωτής ε, έχει θεωρητικά την, επιλογή όταν, αλλάξει όταν αγοράσει ένα αλλατοματικό ε, προϊόν να το επιστρέψει ή να το επισκευάσει. Αλλά μέχρι τώρα ο έμπορος έλεγε, λυπούμε, λοιπόν, το να αντικαταστήσετε αυτό το είδος ε, δεν γίνεται γιατί είναι αμιλητέο το ελάττωμα. Εγώ θα το επισκευάσω. Αυτό λοιπόν που κάναμε για να αποφύγουμε αυτές τις διενέξεις είναι τουλάχιστον να έχουμε ένα ξεκάθαρο κανόνα ότι τουλάχιστον την επιλογή την έχει ο, ο, ο έμπορος και στο μέλλον θα έχει την επιλογή ο έμπερος, αλλά τα πράγματα θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουν θέσει πάρα πολλές αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο. Και εμείς δεν θα αντιταχθούμε να, σε σχέση με την, ως προς την παλαιά διατύπωση του άρθρου 26, να επιστρέψουμε στην παλαιά διατύπωση του άρθρου 26. Ευχαριστώ πολύ μιλάτε για αύξηση στην προσφορά. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούμε για όλους μια ίση ποιότητα, μια ίδια ποιότητα και μια νομική ποιότητα για όλους, κάτι το οποίο δεν είναι πολύ προφανές. Και τώρα κύριε Σβάμπ, σας δίνω, έχετε την τιμή να καταλήξετε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω ότι δεν περιμένετε από μένα να σας απαντήσω όλα τα ερωτήματα. Ε, το είπα άλλωστε και εισαγωγικά αρκετά ξεκάθαρα. Φυσικά δίνω δίκιο σε πολλές ερωτήσεις και νομίζω ότι πολλές ερωτήσεις δεν μπόρεσαν να απαντηθούν σήμερα. Από τη μία επειδή το θέμα αυτό είναι πολύ πλοκό και από την άλλη επειδή δεν έχουμε βρει τις σωστές απαντήσεις. Και γι' αυτό το λόγο εγώ ως εισηγητής θα προσπαθήσω ούτω ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε τι ερωτήσει που μπορούμε να επιλύσουμε και οι ερωτήσει που δεν μπορούν να επιληθούν τελικά να μην εμφανίζονται και στην νομοθεσία. Ωστόσο, θα ήθελα να καταστήσω εξή σαφέ. Εμεί, ω Επιτροπή τη Ιστορική Αγορά ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε νομοθετικό ρόλο. Και δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι εμά δεν μα αρέσει αυτό που έκανε η Επιτροπή, αλλά θα πρέπει στο τέλο να θέσουμε το ερώτημα όχι άμεσα πιο, ποιος βαθμός εναρμόνισης, αλλά ποιο επίπεδο λογικής προστασίας του καταναλωτού. Και αυτό το ερώτημα, σε αυτό το ερώτημα δεν άκουσα σήμερα επαρκής απαντήσεις γιατί όπως είπε η κυρία Τούρμαν, ε, το ερώτημα δεν είναι αν μας αρέσει ο πύχης που θέτει η Κομισιόν όσον αφορά τον καταναλωτή, αλλά το, εμείς θα πρέπει να θέσουμε σε αυτό μας το ερώτημα που εμείς βάζουμε τον πύχη. Και γι' αυτό το θέμα θα πρέπει να συζητήσουμε τους επόμενους μήνες, στο βαθμό που μας το επιτρέπουν οι δυνατότητές μας ε, και ο προπολογισμό μας. Να συζητήσουμε λοιπόν τι θα ήταν πράγματι ένα λογικό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Από πολλές ενώσεις ε, προστασίας των καταναλωτών και από πολλές χώρες λέγεται η οδηγία όσα ε, ε, έχει δεν αξίζει τίποτα, δεν μπορεί να ψηφιστεί. Και ε, βεβαίω εμεί ω Ευρωβουλή μπορούμε να τη βελτιώσουμε σε πολλά σημεία. Και το δύσκολο ερώτημα στο κεφάλαιο 4 είναι κατά πόσο μπορεί κανεί στον ε, τομέα των ε, δικαιωμάτων εγγύηση να ισχύσει εδώ η πλήρη εναρμόνιση. Εδώ υπάρχει, υπάρχουν δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι το συναισθηματικό. Βεβαίω είναι ορθό ότι στο τέλο θα πρέπει να πείσετε του καταναλωτέ ότι αυτό το οποίο αποφασίσαμε είναι ει όφελό του. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Και, αλλά αυτό δεν σημαίνει από τη δική μου σκοπιά ότι σε κάθε σημείο ε, θα πρέπει να πούμε ότι εμείς έχουμε αυξήσει το επίπεδο προστασίας ως προς όλα τα σημεία. Ή για παράδειγμα την τελευταία φορά μιλήσαμε για την ε, προθεσμία ανάκλησης, η επιστροφή του προϊόντος. Ε, εάν είναι 15 μέρες, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να εξηγήσω στους πολίτες ότι μπορούν να αποφελθούν από αυτό. Αλλά εάν υπάρχει μία, αν προβλέπετε ένα διάστημα 10 ετών, είναι δύσκολο να πούμε ότι εάν βάλουμε την περίοδο αυτή, αν παθήσουμε τώρα για αυτό στα 12 χρόνια, αυτό είναι εις του καταναλωτή. Ε, όπως σας είπα, το θέμα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς ε, μπορούμε να πανεύουμε τροπολογίες σε εκείνα τα σημεία της οδηγίας όπου μπορούμε να προωθήσουμε την εσωτερική αγορά, να συμβάλλουμε σε αυτό επικοδομητικά και τελικά να, να σταθμίσουμε ορισμένα τμήματα της οδηγίας και να πούμε ότι εδώ δεν μπορούμε να προβούμε σε μια ενοποίηση. Όσον αφορά όμως τον έλεγχο της εφαρμογής του συσχύοντος δικαίου, εδώ θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί αυτό που σας είπα ήδη εισαγωγικά αφορούσε την ελάχιστη εναρμόνιση, αλλά ακόμα και η ελάχιστη εναρμόνιση δεν τηρείται μέχρι σήμερα. Και ακόμα και εκεί που το επίπεδο δεν είναι ιδεώδες, ακόμα, δεν είναι το ιδανικό, ακόμα και εκεί δεν τηρείται πλήρως. Και σε αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε. Ε, πώς μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα. Επίσης, ε, θα πρέπει να πούμε ότι ίσως κατά περίπτωση υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου η προθεσμία εγγύησης μπορεί ε, ο, μπορεί ο αγοραστής να επιλέξει μεταξύ δύο προϊόντων. Δηλαδή ένα προϊόν έχει μεγαλύτερη διάρκεια εγγύησης και γι' αυτό είναι ακριβό από ένα άλλο προϊόν που έχει μικρότερη εγγύηση αλλά είναι φθηνότερο. Ε, ε, μπορούν δηλαδή να προσαρμοστούν αυτές οι, οι διάρκειες της ε, ανάλογα με το προϊόν και με την περίπτωση. Να υπάρχει μια τέτοια ευελιξία. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωση για την πρόταση της Επιτροπής και υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για την ανταλλαγή απόψεων και για τα επιχειρήματά σας. Ευχαριστούμε κύριε Σβάπ. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε όχι μόνο στο άρθρο 4, σε σχέση όμως με το, τα κεφάλαια 1, 2 και 3 που είχαν εξεταστεί στην Επιτροπή και άλλωστε το Φεβρουάριο η Επιτροπή μας θα διοργανώσει μία, δεύτερη δημόσια ακρόαση στην οποία θα συμμετάσχουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Δηλαδή και εκεί θα έχουμε μία εμπεριστατωμένη ε, ανταλλαγή απόψεων, θα σκεφτούμε με τις χριστουγεννιάτικες αγορές μας στην ε, οδηγία αυτή για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο φάκελο. Παρακαλώ διαθέστε δύο λεφτά σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν θέση. Ça, bonne discussion. Oh, c'était très intéressant, mais la commission est, la commission est dure, hein, Ouh là là. Λοιπόν, θα ξαναξεκινήσουμε για να μπορέσουμε να τελειώσουμε γέρος. Τώρα θα μιλήσουμε για την πολιτική ανταγωνισμού και Προτού δώσω το λόγο στον κύριο Άνταμ Μπίλαν, θα σας δώσω ορισμένες διευκρινήσεις. Να σας πω δηλαδή ότι 19 Νοεμβρίου του 2009 ο πρόεδρος της εσωτερικής αγοράς, ο κύριος Μάικλ Χάρμπορ, που κάθε δίπλα μου έστειλε ε, μία επιστολή στην πρόεδρο της Οικονομικής ε, και Νομισματικής Επιτροπής ζητώντας να καθυστερήσει κατά ένα μήνα την υιοθέτηση της έκθεσης στην ε, ΕΚΟΝ γιατί αυτό θα μας επέτρεπε να έχουμε περισσότερη ευχέρεια και να μπορούμε η έκθεση του κυρίου Μπίλαν ε, να ε, υιοθετηθεί 23 Φεβρουαρίου με ε, ψηφοφορία το Μάρτιο και ολομέλεια, ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Όσοι θέλουν να υποβάλουν όσοι θέλουν να υποβάλουν ε, τροπολογίες πρέπει να το έχουν πράξει μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου, δηλαδή την επόμενη Τετάρτη, άρα πολύ σύντομα και κρατήστε σημείωση. Τώρα όμως κύριε Μπίλαν σας αφήνω το λόγο για να παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβάνουμε ότι 9 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία που έχει καθορίσει η Επιτροπή ΕΚΟΝ. Βεβαίως, εάν θέλουμε να διατυπώσουμε μία γνωμοδότηση, δεν, θα, δεν μας φτάνει αυτός ο χρόνος, διότι ε, πιστεύω ότι η γνωμοδότηση είναι απαραίτηση και γι' αυτό ζητήσαμε να καθυστερήσει η όλη διαδικασία, να πάει δηλαδή ένα μήνα πίσω και ελπίζω ότι η πρόεδρος θα το δεχτεί. Μίλησα με την ε, εκπρόσωπο της γραμματείας, ακόμη δεν έχουμε τελεσίδικη απάντηση, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω η διάσκεψη των προέδρων έχει αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα των ακροάσεων των Επιτροπών και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να το δεχτεί και η Επιτροπή. Τώρα, ε, όσον αφορά την, ε, τη γνωμοδότηση. Όπως είπατε και εσείς σχετικά με την έκθεση ε, για την πολιτική του 2008 η έκθεση αυτή ε, δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο εφέτος. Αποτελείται από έξι ε, κεφάλαια και ένα επιπρόσθετο. Ε, φέτος δηλαδή αποφάσισε η Επιτροπή να προσθέσει ένα κεφάλαιο και αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Τώρα το επιπρόσθετο κεφάλαιο πραγματεύεται τα καρτέλ και τους καταναλωτές. Στο πρώτο κεφάλαιο ε, εξετάζει τις, ε, τους, τους κανονισμούς αντιτράστ ε, στο δύο, πώς χρησιμοποιούνται αυτοί οι κανονισμοί, στο τρίτο εξετάζει τις ενέργειες και δράσεις των ε, καταναλωτών το 2009, το τέσσερα, εξετάζει ε, το, το ευρωπαϊκό δίκτυο ανταγωνισμού. Το 5 και 6 αναφέρεται εις την συνεργασία μεταξύ ε, των θεσμικών οργάνων. Η Επιτροπή ε, ε, ΕΚΟΝ επρόκειτο να εξετάσει την πρώτη έκθεση, το πρώτο σχέδιο της κυρίας ε, Ινβελτ σήμερα. Είχε κατατεθεί το σχέδιο αυτό 20 Νοεμβρίου και νομίζω ότι ε, επηρεάστηκε ιδιαίτερος από το γεγονός ότι το 2008 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά και για την παγκόσμια οικονομία και για την ευρωπαϊκή οικονομία λόγω της σοβαρής κρίσης ε, σε πολλά κράτη-μέλη όπου απεφασίστη να αναλυφθούν ιδιαίτερα μέτρα και δράσεις, να υιοθετηθούν προγράμματα και πακέτα ανακάμψεως και επιπλέον να δοθεί μια ουσιαστική βοήθεια στον τραπεζικό τομέα. Γι' αυτό 11 από τα 21 θέματα στην έκθεση της ε, Επιτροπής ΕΚΟΝ αναφέρονται στις κρατικές ενισχύσεις και στις δράσεις που άπτονται της ε, ε, χρηματο... χρηματικής κρίσεως κατά τη διάρκεια του 2008. Πέραν όμως αυτής της δραστηριότητας θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε έξι σημεία τα οποία πρέπει να ενδιαφέρουν τα μέλη της Επιτροπής σας ιδιαιτέρως. Στο σημείο 2 ο εισηγητής αναφέρεται ε, ε, αναφέρει και προτείνει μία διάταξη για να μπορέσει ε, το Κοινοβούλιο να διαμορφώνει περισσότερο την πολιτική ανταγωνισμού. Στο σημείο 4 ο εισηγητής μας υπενθυμίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού και η αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων είναι πολύ σημαντικές για να λειτουργήσει σωστά η ευρωπαϊκή αγορά και για να προστατεύει το καταναλωτή, άρα δεν νομίζω ότι εδώ πρέπει να έχουμε οποιαδήποτε επιφύλαξη και μετά στο επόμενο κεφάλαιο όσον αφορά την προστασία του ανταγωνισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί τη θέση του σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τις ζημίες και ε, προτείνει ε, να ε, προληφθούν οι μεγάλες αποζημιώσεις για ζημιές. Αυτά όλα είναι θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή μας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις που διατυπώσατε ιδίως ο σκιώδη εισηγητής του ΕΛΚ, ο κύριος Σουάμπ. Το τέταρτο σημείο αναφέρεται στη διάταξη όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί να ενημερώνεται και να προειδοποιείται για οποιαδήποτε αλλαγή η οποία θα αναφέρεται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας κατά τρόπον ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να συμβάλλει και να αναλύει την κατάσταση. Πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντική διάταξη διότι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 ε, όσον αφορά την βιομηχανία, η σχετική διάταξη θα εκπνεύσει το Μάιο του χρόνου άρα η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του θέματος πρέπει να ε, επέλθει πολύ γρήγορα. Στο σημείο 5 λέγεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί να ε, διαβουλεύεται σε οτιδήποτε θέμα συλλογικών εξαιρέσεων από τις συμφωνίες κατά τρόπον ώστε να μπορεί να ελέγχει ικανοποιητικά την κατάσταση και να συμβάλλει. Εδώ πρόκειται ε, πάλι για τις ομαδικές ε, συλλογικές ε, εξαιρέσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και το κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 31 στις ερευνές ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει την έκκληση να εξετάσει την αρχή των δημοσίων διαγωνισμών και να εξετάσει εάν οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών οδηγούν σε μία στρέβλωση του ανταγωνισμού. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά σημεία του σχεδίου της εκθέσεως και ο εισηγητής ε, τονίζει την ανάγκη να υπάρχει μία, ε, μία εξέταση εξ ε, πόστος στις διάφορες χώρες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα διάφορα πακέτα που αναφέρονται στην οικονομία ή στην ανάκαμψη του δημοσίου τομέα. Συμφωνούμε με την αρχή αυτή διότι ουσιαστικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό πρέπει να κάνει, δηλαδή να αξιολογεί ε, τα απλά προγράμματα δραστηριοτήτων. Έχω ε, λάβει σχόλια από τον σκιώδη συγητή του ΕΛΚ θα προσπαθήσω να ενσωματώσω όλα τα σχόλιά του ή στην έκθεση την οποία θα συντάξω. Δεν είχα καιρό να την προετοιμάσω. Ε, δεν πρόκειται να συντάξω πέραν της μία σελίδες και όλα θα γίνουν σε συνεννόηση με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ τον ομιλητή για αυτή την παρουσίαση της έκθεσης και θα δώσω τον λόγο στον κύριο Σοβάμπα γιατί έχει κάποιες παρατηρήσεις για την έκθεση του κύριου Βίλαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Τώρα θα υποφεληθώ ε, από τις συνέργειες γιατί είμαι σκιώδης εισηγητής και στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι η κυρία Ενφέλτ θέλει να επιτύχει κατά, με κάθε τρόπο κοιτάζω αν είναι κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ, ε, να προλάβει την ε, διατηνόμενη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τις ομαδικές απολύσεις. Οπότε γι' αυτό και είμαι διαθέσιμος να παρουσιάσω το ταχύτερο δυνατόν όλες τις τροπολογίες μου διότι είναι ήδη έτοιμες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα αυτό δεν έχει καλύψει πλήρως τις επιπτώσεις ε, της οικονομικής ε, κρίσεως διότι μόνο ελάχιστα ε, μέτρα ελήφθησαν το 2008 για να αποφευθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού στην Ευρώπη και εδώ ενισχύεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα του δικαίωματος ανταγωνισμού και πρέπει εδώ να τονίζουμε τη σημασία του καταναλωτή. Θα αναφερθώ λοιπόν συνοπτικά σε μερικά θέματα τα οποία είναι ενδιαφέρον να συζητήσουμε. Νομίζω ότι στο σημείο που εξετάζουμε πώς θα μπορέσει να εμπλεχθεί περισσότερο ο καταναλωτής ε, για να μπορεί να ε, ζητά αποζημιώσεις ε, για θέματα όπου υφίσταται το ίδιος ζημιά είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει αλλά υπάρχει ο κίνδυνος ότι με αυτόν τον τρόπο θα εκβιάζει κανείς τις επιχειρήσεις και ε, ε, δεν υπάρχει περίπτωση να ε, υπάρξουν μεγάλες αποζημιώσεις στους εργαζόμενους αλλά μεγάλες αμοιβέ στους δικηγόρους που θα υπερασπίζονται τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει το κείμενό της. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε ε, την ε, ε, μεθοδολογία να τρομάξουμε τους επικεφαλείς των μεγάλων καρτέλ διότι σε μια μεγάλη επιχείρηση σαν την Microsoft παραδείγματος χάνει για να αναφέρω μόνο μία βασίζεται εις την ποικιλομορφία των των προϊόντων οπότε τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται είναι σχετικά μικρά αναλογικά ενώ σε μία μικρή επιχείρηση ε, κάποιο, ε, ε, κάποιο πρόστιμο έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο. Πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν καλύτερα στο θέμα των προστήμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, μην τρομάξουν και δεν συμμετάσχουν σε ένα καρτέλ αλλά για να υπάρχει μία ισότιμη μεταχείριση όπως και σε περίπτωση ενός μεγάλου καρτέλ και όχι ε, με χειρότερο τρόπο. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να αναφερθώ στο θέμα της αρχής ανταγωνισμού στα κράτη-μέλη, ε, το one-stop shop όπου ε, μία επιχείρηση τύπου κουαρτέλ ε, μπορεί να αποφύγει ε, τις, τις δηλώσεως του τι, πώς λειτουργεί αλλά αν το αποφύγει σε μία χώρα δεν θα μπορέσει να το επιτύχει παντού και γι' αυτό θα πρέπει να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εδώ για το, η Μεγάλη Βρετανία παραδείγματο χάρη ε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και θε, περιμένω να δω πόσο σκοπεύει ε, να διατηρήσει το αποτρεπτικό αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κείμενό της εδώ δεν αναφερόμαστε μόνο στους καταναλωτές αλλά και σε ορισμένες επιχειρήσεις στις οποίες επευλήθηκαν πρόστιμα και πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει και να μας ενημερώσει καταρχήν εάν ε, τα ε, προγράμματα των κρατών μελών μπόρεσαν αποτελεσματικά να ε, αντεπεξέλθουν της οικονομικής κρίσεως, τι, τι πόροι διατέθηκαν και ούτω καθεξής και επίσης αν υπάρχουν επιχειρήσεις με προεξέχουσα θέση τις οποίες θα πρέπει να καταπολεμήσουμε. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Στήλερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον, εισηγη... εισηγητή και τον σκιώδη εισηγητή για τη συμβολή τους. Νομίζω πως είναι σημαντικό το ότι γίνεται λόγος για λιγότερα καρτέλ. Εγώ δεν είχα ιδέα πώς επηρεάζονται όλα αυτά τα μένα από τα δύο. Πολλά προϊόντα ε, θίγονται εδώ, αλλά και θέματα τα οποία ποτέ δεν θα σκεφτόμασταν ε, είχαν επιπτώσεις ε, για τους ίδιους μας τους εκλογές. Εγώ είμαι αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Οίκων και με την έκθεση άκουσε άκουσα ήδη τα σχετικά πράγματα. Προσπαθεί να τα πει όλα εμπεριστατωμένα. Ο κύριος Βάμπ μίλησε για τη, την ψηφιακή και την ηλεκτρονική επικοινωνία. Στη σελίδα 20 μιλά για όλα αυτά και έχει ένα σημαντικό σημείο το 16 στη σελίδα 20 όπου λέει για τη διαθεσιμότητα της ευρεία και στο 17 μιλά για την επόμενη γενεά και την πρόσβαση στα δίκτυα τα ευρυζωνικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό συζητούσαμε και προηγουμένως, ότι κανένας δεν πρέπει να μείνει πίσω. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Ο προηγούμενος ομιλητής μίλησε για την Microsoft, την Intel, υπήρχε και το θέμα των ευκαιριών και των φραγμών online και για το σχέδιο της συνολικής εξαίρεσης που αναφέρεται στο σημείο 24 της ε, κυρίας Σιντφέλτ και 25 και ίσως η Κομισιόν εδώ μπορεί να βοηθήσει. Αλλά σελίδα 24, σελίδα 19, στην παράγραφο 19, συγγνώμη, στην προτελευταία πρόταση γίνεται λόγος που είναι ιδιαίτερα προσφυλές στους δικούς μου ε, συμπολίτες Δηλαδή την έρευνα για την Κάρπαρ και την Northlink, και από ό,τι κατάλαβα ολοκληρώθηκε η έρευνα την περασμένη εβδομάδα, αλλά οι ευρωβουλευτέ δεν πήραν τίποτα πληροφορία σχετικά. Οι Σκοτσέζοι, μάλιστα, ευρωβουλευτέ δεν ενημερώθηκαν. Από ό,τι κατάλαβα δεν υπήρξε ρήξη των κανόνων ανταγωνισμού, ότι η Σκοτσέζικη κυβέρνηση είχε συμμορφωθεί προ του κανόνε αυτού, αλλά εν πάση περιπτώσει θα εκτιμούσαμε να μα στείλει τι σχετικέ πληροφορίε η Κομισιόν για τη φαρμακοβιομηχανία. Πολύ σημαντικό σημείο για τους καταναλωτές και στη δική μας έκθεση θα έπρεπε να αναφέρουμε τη σημασία αυτής της βιομηχανίας. Ε, νομίζω πως ε, έγινε ήδη λόγος γι' αυτό. Και τέλος. Κάτι που η Σόφη Ιντεφελτ έχει πει στη σελίδα 13 για την πράσινη οικονομία και την πράσινη ανάκαμψη. Ε, πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς γίνεται λόγος για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Είναι μεγάλο άρθρο για τις πράσινες θέσεις, την πράσινη ε, εργασία και τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τον Σκιώδη. Και... και είμαι βεβαία ότι θα έχουμε ε, καλή συνεργασία και είναι πολύ σημαντικό να ε, βρούμε μια σωστή συμφωνία. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρούλα ζήτησε το λόγο. Όχι. Κύριε Χάρμπορ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Καταρχήν, όπως όλοι τόνισαν, η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο για τις επιπτώσεις του καταναλωτή σε περιπτώσει ανταγωνισμού, πράγμα το οποίο αιτιολογεί τη σύνταξη γνωμοδότηση προ την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Ελπίζω πω θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, επιτυχώς. Επίσης, έχουμε ίσως το πλονέκτημα, γιατί η κυρία Ιντβέλτ έχει ήδη συντάξει την έκθεσή της και άρα μπορούμε να δούμε τους τομείς όπου θα μπορούσε να συμβάλλει η Επιτροπή μας και θα πρέπει αυτό να το εξετάσουμε ε, προσεκτικά. Δεύτερη παρατήρηση είναι αυτό το σχόλιο που φορά τα είναι συνολική εξαίρεση για τα οχήματα με κινητήρα. Εμείς ε, ζητήσαμε να συμμετέχουμε, γιατί υπήρχαν διάφορα θέματα, ιδιαίτερα για τις επισκευές οχημάτων. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ανταγωνισμού ε, ετοιμάζει ένα νέο κανονισμό επ' αυτού και είναι σωστό να ζητήσουμε να έχουμε χρόνο για να το εξετάσουμε, ακόμα και αν δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε αυτή την επιχείρηση, γιατί θέλουμε τα ωφέλη για τους καταναλωτές σύντομα. Αλλά ορισμένοι από εσά ε, έχουν ενημερωθεί από τον ε, κλάδο των επισκευαστών να το καθυστερήσουν. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ε, καταστεί ισχύουσα όσο γίνεται πιο σύντομα. κάναμε και ακρόαση για το, την συνολική αυτή εξαίρεση και φαίνεται να θέλουν να το περάσουν τελευταία στιγμή και αυτό είναι σημαντικό. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για την Επιτροπή μας. Ιδιαίτερα έχει να κάνει με τι, τα θέματα ε, για τα αγαθά συγκεκριμένου σήματος. Ε, Τελευταία μου παρατήρηση είναι ότι η κυρία Ιντβελτ και ο κύριος Βίλεν ε, ανέφεραν το θέμα των, των δημοσίων προμηθειών που σαφώς είναι δικό μας θέμα, δική μας ευθύνη και από ό,τι κατάλαβα, η έκθεση της κυρίας Σίντφελτ ζητά διερεύνηση για την εφαρμογή των κανόνων γενική ε, δημοσίων προμηθειών. Ίσως η Κομισιόν θα μπορούσε αυτό να το επιβεβαιώσει. Νομίζω πως υπάρχουν πτυχές των δημοσίων προμηθειών όπου ισχύουν οι κανόνες ανταγωνισμού, αλλά νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε σαφείς πως αυτό είναι δική μας ευθύνη και η κυρία Ρούλε ακριβώς αυτά τα θέματα διερευνά. Πάντω σαφώς μπορούμε να δούμε από τη σύντομη συζήτηση πως υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη και μπορείτε να βασιστείτε σε μένα ότι θα υπερασπίσει το δικαίωμά μας να το κάνουμε αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η κυρία Ρούλε έχει το λόγο. Που σίγουρα θα μιλήσει για τις δημόσιες προμήθειες. Ευχαριστώ. Σχετικά με, τις, ε, ε, με τους δημόσιους διαγωνισμούς. Ε, υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν επικαλύπτεται καθόλου και καλύπτει νέα προβλήματα, δηλαδή ότι υπάρχουν κράτη, κρατικές εταιρείες οι οποίες προσέρχονται στην κρατική αγορά και εάν αυτές βοηθούν ε, τις ε, δικές τους επιχειρήσεις χωρίς να συμμορφώνονται εις ε, την απαγόρευση κρατικών ενισχύσεων που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουμε προβλήματα και για τον οικοδομικό τομέα και ε, για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και για, την, και για τις οικοδομές όπως ήδη σας είπα. Αλλά με τα θέματα αυτά πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο περισσότερο η Επιτροπή Ίντα. Δηλαδή, εάν υπάρχει διαφορετική εφαρμογή οδηγιών σε διάφορα κράτη-μέλη που οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού, θα πρέπει να το εξετάσουμε. Δεν ξέρω όμως, ε, θα έπρεπε να ρωτήσουμε ίσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, διότι βλέπουμε συνέχεια ότι μία οδηγία ε, εφαρμόζεται διαφορετικά διαφορετικά από το ένα κράτος στο άλλο και αυτό το οποίο με ενδιαφέρει για τις ε, δημόσιες προμήθειες και τους δημόσιους διαγωνισμούς είναι να επιτύχουμε μεγαλύτερη νομική ασφάλεια διότι όταν η τοπική αυτοδιοίκηση, ιδίω η μικρή τοπική αυτοδιοίκηση ε, αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα τότε το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί και από όλους τους τομείς της οικονομίας. Σας ευχαριστώ. Νομίζω πως θα τώρα καλό να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που την αντιπροσωπεύει η κυρία Κουλούτσι. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την απόψινή συζήτηση γιατί μας έδωσε μια συνολική εικόνα για τα ενδιαφέροντα της Επιτροπής και μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την ε, κτίσια έκθεση για τον ανταγωνισμό και να ξεκινήσουμε ένα καλό διάλογο που θα μας επιτρέπει να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα. Επίσης, θα ήθελα να θυμίσω, και το γνωρίζετε αυτό ήδη, είναι ότι φυσικά είμαστε εμείς ε, οι διεκπαιρεωτές στην Κομισιόν και οι μόνοι ε, μάλλον είμαστε σε μια ενδιάμεση κατάσταση σε σχέση με την Κομισιόν, όπως γνωρίζετε, και δεν μπορώ να σας δώσω υπεύθυνες απαντήσεις. Θα είμαι κάπως ε, προσεκτική στις σημερινές απόψινές μου απαντήσεις, γιατί δεν μπορώ να ε, δεσμευτώ για την επόμενη Επιτροπή. Ε, το θέμα των ε, κρατικών προμηθειών, ε, ναι, είναι όντως είναι περισσότερο αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, και, αλλά εννοείται ότι η στρέβλωση ανταγωνισμού, αν συμβεί σε κρατικές προμήθειες, θα το εξετάσουμε εμείς, αλλά όχι στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αυτή τη στιγμή μελετάμε. Συζητάμε, λοιπόν, αλλά ο βασικός κανονισμός σχετικά με τα θέματα αυτά ανήκει στην ΓΔ αγορά. Για τον δίκαιο ανταγωνισμό, το θεμητό ανταγωνισμό, ακούσατε πως υπήρξαν αλλαγές στις αρμοδιότητες της ΓΔ ανταγωνισμού, γιατί θα ασχοληθούμε με τις κρατικές ενισχύσεις των τομέα των μεταφορών. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα αλλά θα, σας θα ενημερωθούμε και θα επανέλθουμε για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Καλωσορίζουμε το ενδιαφέρον που έχετε λοιπόν για όλα αυτά τα θέματα. Μπορώ να σας πω ότι προσπαθούμε να ενημερώνουμε το Κοινοβούλιο για τη συζήτηση και τη δημόσια διαβούλευση στην οποία αναφερθήκατε. Ήταν μια πολύ καλ... ένα πολύ καλό εγχείρημα και το εργαστήριο και νομίζω πως βοήθησε στη συζήτηση. Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για να ανταλλάξουμε απόψεις από αυτού και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να λάβουμε υπόψη τα σχόλιά σας. Θα πρέπει να σας θυμίσω παρ' αυτά ότι ο κανονισμός για τη συνολική εξαίρεση θα εκπνεύσει τον Μάιο, οπότε δεσμευόμαστε από κάποιους νομικούς περιορισμούς, αλλά και πάλι επαναλαμβάνω, καλωσορίζουμε τα σχόλια και προσπαθούμε να τα λάβουμε υπόψη όσο γίνεται περισσότερο. Η ΕΚΟΝ Πραγματικά θα πρέπει να ε, ακολουθήσει το γενικό χρονοδιάγραμμα. Η έμφαση που δίνουμε στους καταναλωτές στην έκθεσή μας είναι κάτι το οποίο θεωρούμε πολύ σημαντικό και εκτιμούμε που η Επιτροπή σας αναγνωρίζει αυτή την πτυχή. Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε λοιπόν φέτος και θα το επαναλάβουμε και τα επόμενα χρόνια καθώς θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τα πιο σημαντικά θέματα σημεία του ανταγωνισμού και να τα εξηγήσουμε με όσο γίνεται πιο παιδαγωγικό τρόπο και στους καταναλωτές. περισσότεροι τόνισαν ε, ότι το 2008 αφορούσε περισσότερο την ε, χρηματοπιστωτική κρίση και είμαστε ευγνώμονες για τα σχόλια που ακούσαμε σήμερα. Για το πιο συγκεκριμένο θέμα των ε, ιδιωτικών ζημιών ή βλαβών, ακούσαμε με ενδιαφέρον τα σχόλια του κύριου Σβάμπ και θα προσέχουμε. Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε και περαιτέρω σχόλια και συζήτηση. Ευχαριστούμε κύριε Κολούτσι. Κύριε Βίλαν, έχετε κάτι να προσθέσετε σύντομα. Ναι. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Μας μένουν μόνο πέντε λεπτά. Θα ήθελα να πω ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. <coughs> για την ε, συνεργασία τους. Σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε Ε, και εκείνους που συμμετέχουν και στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ε, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Χάρμπορ γιατί τόνισε ότι θα αγωνιστεί ώστε να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότησή μας στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Κάτι το οποίο ανέφερα και εγώ στι αρχικέ μου παρατηρήσει. Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, ένα από τα έξι κεφάλαια τη έκθεση ΕΚΟΝ, το οποίο είναι αφιερωμένο σε θέματα καταναλωτή και προφανώς και σαφώς θα πρέπει να συνοδεύεται η έκθεση αυτή από δική μας νομοδότηση. Και επίσης το θέμα της δημόσιας ε, των κρατικών προμηθειών αναφέρθηκε. Η κυρία Ρούλε αναφέρθηκε σε κάτι που αφορά και την Πολωνία, κινέζικες εταιρείες και εταιρείες από άλλες χώρες, αλλά ιδιαίτερα κινέζικες εταιρείες που λαμβάνουν κρατική βοήθεια και με αυτόν τον τρόπο παραβιάζουν τις αρχές του ανταγωνισμού. Αλλά αυτό είναι κάτι επί το οποίο θα πρέπει να δουλέψει η Επιτροπή Σα ευχαριστώ και πάλι για τι παρατηρήσει σα και ελπίζω πω θα είμαστε σε θέση να δουλέψουμε αποτελεσματικά για αυτή τη γνωμοδότηση. Σα ευχαριστώ. Τελευταία παρατήρηση. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ΙΜΚΟ θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου στις 18.30 στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ για αυτές τις επικοδομητικές συζητήσεις και θα δώσω το λόγο στον κύριο Προεδρό για να κλείσει τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω που προεδρεύσατε τόσο καλά απόψε και όλους τους αντιπρόεδρους επίσης, γιατί νομίζω ότι είναι ε, προφανώς ότι μοιραζόμαστε τη δουλειά της Επιτροπής. Και αυτό γιατί δεν θα έχουμε πλήρη συνεδρίαση μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, 25 Ιανουαρίου, πολύ καιρό από τώρα δηλαδή, λόγω του χρονοδιαγράμματος και με τις ακροάσεις επίσης που έχουμε ενδιάμεσα. Ε, πάντως, σε περίπτωση που δεν σας δω, σας εύχομαι... Ε, Ό,τι καλύτερο για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Ελπίζω να ξεκουραστείτε κιόλας. Ξέρω πως ορισμένοι συγκητές θα πρέπει να συντάξουν τις εκθέσεις τους και σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας σε εμένα στους τρεις πρώτους μήνες εργασίας ως Πρόεδρου γιατί πιστεύω πως κάναμε καλή αρχή, είχαμε πλήρη ημερήσια διάταξη και δεν αφήσαμε να μας καθυστερήσει η μεταβατική περίοδος για την ε, Επιτροπή. Πιστεύω πως θα είναι καλό θεμέλιο για αποτελεσματικότητα και το 2010. Σας ευχαριστώ, καλό σας βράδυ και ευχαριστώ και πάλι την Περναντέτ. Αν στο Στρασβούργο για τη συνάντηση με τον καθηγητή Μόντι.